Καλημέρα σας. Ξεκινούμε και πάλι τις συζητήσεις μας. Σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη με τη γνωμοδότηση του συναδέλφου κυρίου Βόρνα για την πολιτική της συνοχής στη Βόρεια Ιρλανδία. Ελπίζω να έχετε μαζί τις κάρτες για την ψηφοφορία γιατί ξεκινούμε αμέσως. Ο συνάδελφος είναι εδώ. Εάν είσαστε όλοι λοιπόν έτοιμοι μπορώ να ξεκινήσω. Με την τροπολογία 3 υπέρ. Μάλιστα. Ε, έχετε αντιρρήσεις ε, να ψηφίσουμε όλοι on block. Όχι. Αντιρρήσεις όχι. Λοιπόν ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες ομού. Ηλεκτρονικά, αν θέλετε, αρχίζει η ψηφοφορία. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 11. Υπέρ με ψήφο κατά και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνούμε στο σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως με το κλασικό πρόβλημα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα ε, χρονικά περιθώρια για, την, ε, για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Βεβαίως αυτό απασχολεί και το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όχι μόνο εμάς, αλλά πρέπει να συντομεύσουμε τις ε, περιόδους. Συνήθως έχουμε μια έκθεση που δημοσιεύεται Οκτώβριο-Νοέμβριο, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως και από το Συμβούλιο υπάρχει πρόβλημα, γιατί δίνουμε απαλλαγή με βάση σύσταση του Συμβουλίου. Και αν δεν υπάρχει αυτή η σύσταση, τυπικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα το Συμβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό πρόσκομα στην προσπάθεια για συντόμευση των χρόνων. Και βεβαίως θέλουμε πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε τα θέματα σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ταυτόχρονα και να καλέσουμε όλους τους ενδιαφερομένους σε μία συζήτηση Και βεβαίως η Επιτροπή πάλι εξαρτάται για την υποβολή των δικών της ε, ε, εκθέσεων από την υποβολή των λογαριασμών των κρατών μελών. Κλασική ιστορία, πολλές φορές την έχουμε αντιμετωπίσει χρόνια τώρα και προσπαθούμε και από τις ομάδες εργασίας να βρούμε λύσεις συντομεύοντας τους χρόνους και τα χρονοδιογράμματα. Ξέρουμε ότι δεν, δεν έχουμε γίνει πολύ αγαπητοί γι' αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Χαίρομαι για την παρουσία του ελεγκτικού συνεδρίου εδώ και του δίνω μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Γκρέκο, παρακαλώ. Το μικρόφωνο του ομιλητή, παρακαλώ. Ωραία, βρήκα το σωστό κουμπί. Καλημέρα σας, λέει ο κύριος Γκρέγκορ και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε, που έχετε προσκαλέσει το ελεκτικό συνέδριο για την τόσο σημαντική αυτή συζήτηση. Σημειώνω ότι μας έχει απασχολήσει πολύ το θέμα της συντόμευσης των χρόνων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας και έχω και στοιχεία ούτως υπήν για το πόσο μας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό. Παραδείγματι έχουμε σκεφτεί από τα μέσα Νοεμβρίου να μεταθέσουμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου αρχάς ε, Οκτωβρίου την υποβολή της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου τα τελευταία χρόνια. Έχουμε επίσης αναλύσει διεξοδικά τις προθεσμίες σε σχέση με, τους το δημοσιονομικό κανονισμό. Το έχουμε περιγράψει αυτό σε γνωμοδότησή μας. Δηλαδή προτείνουμε πιο σύντομα ε, προθεσμίες για τα διάφορα έγγραφα, για την κατάθεση των διαφορών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ε, απολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε επίσης να βρούμε λύσεις σε σχέση με, τις, ε, με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, των οποίων επίσης καθυστερούν συχνά οι ισολογισμοί και βέβαια πρέπει να κατατίθενται 1η Οκτωβρίου με βάση τους ε, κανόνες οι σχετικές εκθέσεις από πλευράς μας Ετοιμάσαμε πέρσι ε, μια περιληπτική έκθεση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς μέσα στην ετήσια έκθεση και για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για τον έλεγχο του 2017, ετοιμάζουμε μία έκθεση και για τους 41 και όχι 41 ειδικέ εκθέσεις για κάθε ε, αποκεντρωμένο οργανισμό, μία δηλαδή. Έτσι λοιπόν με τη συγκέντρωση αυτή των εκθέσεων σε ένα έγγραφο ίσως μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της απαλλαγής. Βέβαια παραμένουν κάποια στοιχεία που εμποδίζουν περαιτέρω πρόοδο και στο μευσή των προθεσμίων. Καταρχάς ότι η δική μας η εξέταση των ε, ισολογισμών στηρίζεται σε ενοποιημένους ετήσιους ισολογισμούς, πράγμα το οποίο μας δεσμεύει. Και βέβαια έχουμε και τον έλεγχο της νομιμότητας στα κοινά τμήματα. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία από πλευρά τη Επιτροπή που φαντάζομαι θα σχολιάσουν οι συνάδελφοι τη Επιτροπής. Εγώ ήθελα απλώ να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί νωρίτερα από τον Μάιο που τελικά προτείνεται το έγγραφο το σχετικό με, τις, ε, με, το παθητικό, με τα παθητικά. Εν ολίγης πρέπει βεβαίως και να γίνουν οι μεταφράσεις σε επίσημες ε, γλώσσες, ε, όπου βέβαια ο καταλληλότερος χρόνος είναι ο Αύγουστος, καταλληλότερος μήνας, κατά τον οποίον κάνουμε τη δική μας την προσπάθεια για, τη, για την καλή μετάφραση της ετήσιας έκθεσης. Φυσικά, να πάσα στιγμή είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε νέες προσαρμογές των ε, χρονοδιαγραμμάτων, αλλά πρέπει ότι αποφασιστεί να είναι και εφικτό και ρεαλιστικό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε λογικά να δεσμευτούμε να καταθέτουμε ε, μία-δύο εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου την έκθεση, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από, την, ε, από τις λοιπές ε, προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα και από την καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Και πάντα το κέριο ζήτημα θα είναι το πώς θα γίνει η εξέταση των ισολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Επίση, η στρατηγική του ερευνητικού συνεδρίου είναι τριετή. Έχουμε αναλογιστεί τη δυνατότητα βελτίωσης ε, της ε, ποιότητας. Έτσι λοιπόν ναι, δίνουμε μια έκθεση αιτήσεων επιδόσεων ε, που θα μπορούσε να δημοσιεύεται στα αρχά Ιουνίου και αυτό μπορεί νομίζω να συζητηθεί στη σημερινή σας ε, ανταλλαγή απόψεων. Ίσως μια άλλη λύση θα ήταν ένα κομμάτι συγκεκριμένο της ετήσιας έκθεσης να κατατίθεται το Νοέμβριο. Και έτσι θα μπορούσατε και εσείς αλλά και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς να ε, είναι εν γνώση αλλά αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα, μας θα σας απασχολήσει στην προσεχή ε, απαλλαγή. με βάση και τη γνωμοδότηση και, την, ε, και τον απολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε σε θέση σας για να απαντήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρέγκορ δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ ικανοποιημένη. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε ή τι πρέπει να γίνει για να μπορεί να καταθέτει το ελεγκτικό συνέδριο την ε, έκθεση του τον Ιούνιο, πριν από τις θερινές διακοπές δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Κύριος Γκρέγκορ, ναι, όπως είπα ακροφυγός, εξαρτώμεθα από τα έγγραφα που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως ένα στοιχείο θα ήταν η Επιτροπή να καταθέτει τους ισολογισμούς ε, στη, την 1η Μαρτίου και να έχουμε ενοποιημένους τελικούς ισολογισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου μετά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μετακυλείται ο φόρτος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, όπως είπα, Αντί για 41 ειδικέ εκθέσεις σκεφτόμαστε να δημοσιεύουμε μία ενοποιημένη και για, τις 40, για τους 41 αποκεντρωμένους οργανισμούς, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα λαμβάνουμε τους ε, δημοσιονομικούς ισολογισμούς των ε, υπηρεσιών που μέχρι τώρα κατατίθενται 1η Αυγούστου. Αν αυτό μπορεί να έρθει πιο νωρίς, τότε και εμείς μπορούμε να τελειώνουμε νωρίτερα αυτή την ενοποιημένη έκθεση η Πρόεδρος. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει πρόβλημα για τους ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς να καταθέτουν νωρίτερα τους ε, ισολογισμούς έτσι ώστε να διευκολύνουν ε, την διεξαγωγή της διαδικασίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε εκπρόσωπους, εκπρόσωπο και πολλών αποκεντρωμένων οργανισμών. κυρία Τούλης παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Από το δίκτυο των ε, ε, εξωτερικών υπηρεσιών και εμείς είμαστε υπέρ της προώθησης της διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής. Αλλά όπως είπατε και εισαγωγικά, έχουμε πολλούς διάφορους ε, φορείς που εμπλέκονται και εμείς είμαστε πιο πολύ από την πλευρά της αντίδρασης και όχι τόσο πολύ από την πλευρά της δράσης. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν λάβουμε τα σχετικά έγγραφα με τις παρατηρήσεις του, δικαστηρίου, του Ελληνικού Συνεδρίου ή το αριθμοτολόγιο του Κοινοβουλίου. Όσο τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και να προωθήσουμε τη διαδικασία της απαλλαγής. Ένα μόνο θέμα θα θέλω να σας επισημάνω. Συνήθως οι υπηρεσίες, οι Εξαιρετικές αυτές ε, υπηρεσίες ε, των οργανισμών που είναι υπεύθυνε για το κλείσιμο του έτους, είναι αυτές που είναι υπεύθυνε και για τη χορήγηση της απαλλαγής. Άρα αυτό σημαίνει διπλή δουλειά για αυτές τις υπηρεσίες και υπεβάρυνση για τις ε, υπηρεσίες αυτές. Αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε άρεστοι στην ποιότητα όπως είμαστε και στο παρελθόν. Να σας κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Τι εννοείτε ότι είστε πρόθυμοι και υπάρχει βούληση. Τι αντίσταση ενδεχομένω να υπάρξει. Μπορούμε λοιπόν να ε, επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή τον Απρίλιο, να λαμβάνει όλα τα στοιχεία, το ελεκτικό συνείδριο, τα στοιχεία αυτά τον Απρίλιο. Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφορά, είναι μόνο διαδικαστικές, ε, διαδικαστικά ζητήματα. Όπως ξέρετε, έχουμε και τις εταιρείες ε, διεξαγωγής ε, ελέγχου η τρέχουσα λοιπόν προθεσμία είναι η 1η Αυγούστου και οι εξωτερικέ υπηρεσίε χρησιμοποιούν μία σύμβαση πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει αυτός ο οικονομικός έλεγχος. Εδώ λοιπόν μπορούμε να παρέμβουμε σε ό,τι αφορά την υποβολή αυτή της έκθεσης. Δεν μπορώ να μιλήσω από πλευράς του Ελληνικού Συνεδρίου τι θα χρειαζόταν δηλαδή το ηλεκτρικό συνέδριο προκειμένου να υπάρξει ο συντονισμό μεταξύ των, των εταιριών εξωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών ελεκτών. Γιατί όλο το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στη σύμβαση πλαίσιο λίγο πολύ αναφέρει τι θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι πότε. Εγώ μιλώ για τη Frontex για παράδειγμα. Έχουμε τους εξωτερικού ελεγκτές που κάνουν τον έλεγχο τον Φεβρουάριο και μετά τον Ιούνιο για μια δεύτερη επίσκεψη. Αυτό μπορούμε να το μετατοπίσουμε χρονικά, να το βάλουμε πιο νωρί. Να το συζητήσουμε, αλλά σε τελική ανάλυση θα πρέπει να τροποποιηθεί και αυτή η σύμβαση πλαίσιο. Και στη συνέχεια για τα ερωτηματολόγια. Έχουμε διάφορα ερωτηματολόγια. Και έχουμε συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο προκειμένου να είναι τυποποιημένο το ερωτηματολόγιο αυτό για όλα τα, όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες. Γιατί ξέρετε, όσο πιο τυποποιημένα είναι τα ερωτηματολόγια, τόσο πιο εύκολο και γρήγορο είναι το έργο της συμπλήρωσής τους. Και έτσι είμαστε στην ώρα μας. Το αρτηματολόγιο, αν κατάλαβα σωστά, θα το συζητήσετε σήμερα. Αν ε, το λάβουμε άμεσα την επόμενη εβδομάδα, θα σας ε, υποβάλλουμε τις σχετικές απαντήσεις μέχρι τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει θέμα. Και στη συνέχεια υπάρχει η σύνδεση αυτή και θα θέλαμε να ξανακάνουμε την πρόταση που έχουμε κάνει στο παρελθόν προκειμένου το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο να ενσωματωθεί με τις ερωτήσεις ε, και τα σχόλια για τις προηγούμενες ε, απαλλαγές. Υπάρχουν επίσης ε, και οι μεμονωμένες ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται μετά την υποβολή της έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου. Αν δημοσιεύονται λοιπόν πιο νωρίς οι εκθέσεις του Ελληνικού Συνεδρίου, μπορούν να αποστέλλονται και πιο νωρί στο δίκτυο των εξωτερικών υπηρεσιών και Και μέσα σε τρεις εβδομάδες ε, θα κάνουμε τη σχετική μελέτη για να μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα ενοποιημένο κείμενο στις αρχές χορηγήσης της απαλλαγής. Ευχαριστώ. Yeah. ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τα βλέμματα στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς ε, Λοιπόν, θα μας πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ημερομηνία αυτή για την 1η Αυγούστου, το ελεκτικό συνέδριο. Ε, μπορούμε να καθορίσουμε έτσι το πρόγραμμά μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη διαδικασία αυτή. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και από μας εξαρτάται στην τελική ανάλυση. Έχετε το λόγο. Ναι, βεβαίω μπορούμε να συνεργαστούμε με όλους όσους πήραν το λόγο για να βρούμε κάποιους τρόπους για να βελτιώσουμε τους ρυθμούς ε, ε, αυτών των εκθέσεων αλλά θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλίζει μια ποιοτική διαδικασία ε, σε, όλες τις, σε όλα τα στάδια. Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε τμηματικά. Φέτος δηλαδή να επιταχύνουμε κάπως τη διαδικασία, αλλά να συζητήσουμε επίσης και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πού βρισκόμαστε φέτος. Παρουσιάσαμε στο ελεγκτικό συνέδριο και καταθέσαμε τους προσωρινούς λογαριασμούς. Ε, σύντομα ε, θα κλείσει ε, το σχέδιο ελέγχου. Ε, και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ε, εγκρίνουμε το τελικό σχέδιο έτσι ώστε να εγκριθούν οι ενοποιημένοι λογαριασμοί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η έκθεση για την ετήσια διαχείριση 15 ε, Ιουνίου θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου ως έκθεση απόδοσης η έκθεση για την απόδοση ε, μέσα Ιουνίου και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί τέλη Ιουνίου, έτσι ώστε να έχετε το χρόνο να συζητήσετε τα διάφορα έγγραφα. Τώρα, για τους εξωτερικούς οργανισμούς και την σύμβαση πλαίσιο, θέλω να το κοιτάξω σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν έχω εδώ όλες τις πληροφορίες, αλλά... Ε, είμαι υπεύθυνη για κάποιους από αυτούς τους οργανισμούς και έχω λάβει ε, feedback από τους εξωτερικούς ελεγκτές και με τον τρόπο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την απόκρισή τους, ε, έχω να σας πω πως τα τελικά στοιχεία θα τα έχουμε μόνο τέλη Αυγούστου, αλλά θα δω στην ε, σύμβαση πλαίσιο αν χρειάζεται κάποια τροποποίηση. Πάντως κάθε χρόνο, κάθε οργανισμός υπογράφει μια συγκεκριμένη ε, σύμβαση με μια ελεγκτική εταιρεία και τότε στη στιγμή αυτή θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των αποτελεσμάτων ελέγχου. Αυτά είχα να σας πω και ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για να συζητήσουμε μακροπρόθεσμα ποια θα ήταν τα στάδια έτσι ώστε να κάνουμε κάτι για να είναι πιο σύντομη η όλη διαδικασία. Ναι, ευχαριστώ. Έτσι το είχα σκεφτεί και εγώ. Όλοι να δείξουν καλή διάθεση μεν, αλλά αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βγάλουμε δεν. Ας μην ε, χάσουμε λοιπόν το στόχο μας, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πολύ ωραίο να κάνουν όλη την προσπάθειά τους, αλλά δεν αρκεί η προσπάθεια σε αυτήν την περίπτωση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, πάνω απ' όλα, τα κράτη-μέλη και τα δεδομένα ε, που σας ε, καταθέτουν για να κάνετε εσείς τις εκθέσεις προς το ελεγκτικό συνέδριο, τι ρόλο παίζουν, σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την όλη διαδικασία και βέβαια το εγχείρημα της ε, περικοπής των χρόνων στην ε, εκτέλεση του προπολογισμού. Γιατί δεν είμαι πολύ ε, αισιόδοξη σε σχέση με τα κρατημέλη, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουμε ποτέ παρόντα από το Συμβούλιο ή υπάρχει κανείς εδώ τυχαία, όχι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Συμβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει πιο μπροστά τις διαδικασίες. Είναι η ίδια ομάδα εργασίας τελευταία ανάλυση, αυτή που ασχολείται με τον προϋπολογισμό και μετά με την απαλλαγή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άντρες όπως και να έχει δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά με το multitasking και για τις γυναίκες δεν είναι βέβαιο και αυτό καλό θα ήταν να υπάρχει μια διαφορετική σύνθεση. Ε, το Φεβρουάριο έχουμε ένα κατάλογο με τις συστάσεις του Συμβουλίου και για τον τύπο βέβαια περιμένει το Κοινοβούλιο η Ολομέλεια για να ε, λάβει τις αποφάσεις του αλλά το χρόνο νομίζω θα προλαβαίνουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Θα λαμβάνουμε αποφάσεις δηλαδή πριν από το Συμβούλιο. Θα προκύψουν οπωσδήποτε ε, συγκρούσεις και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα βγει, αλλά εγώ είμαι διατεθειμένη να περικόψω τη διαδικασία, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθυστερούμε τόσο πολύ. Και μετά ας δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο, αν εμείς περικόψουμε από τη δική μας πλευρά τη διαδικασία, τους χρόνους της απαλλαγής. Και όταν ξέρουμε το Συμβούλιο δεν πηγαίνει και τόσο εις βάθος όσο εμείς. Ε, εν πάση περιπτώσει, βέβαια, είναι σημαντικέ ε, οι θέσει του Συμβουλίου σε αυτό. Κοιτάξτε εσεί από την Επιτροπή, παρακαλώ, να μα πείτε λίγο περισσότερο τι ρόλο έχουν τα κράτη-μέλη και τι δυνατότητε βλέπετε για ε, περικοπή των ε, χρόνων. Και εσεί, κύριε Γκρέγκορ, πείτε μα στη διάρκεια του χρόνου ποιες εργασίες ε, πότε ολοκληρώνονται, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή τη διαδικασία ε, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, με την ενοποιημένη έκθεση όπως είπατε και τι άλλες δυνατότητες βλέπετε για περιορισμό. Και βέβαια και εμείς από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας πιο βιαστικά, πιο γρήγορα. Ε, κύριε Γκρέγκορ, πότε είναι έτοιμη για να πάει στη μετάφραση η έκθεση. τη Φερρυπίν θα μπορούσαμε ένα μέρος της δουλειάς να το διευθετούσαμε με ένα προκαταρκτικό σχέδιο, με ένα πρώτο σχέδιο το ΣΥΠΗΝ, χωρίς να περιμένουμε τη μετάφραση όλες τις γλώσσες. Δεν ξέρω αν εδώ ε, παραβιάζω διάφορα ταμπού και ιερά, ιερές αρχές, αλλά μήπως ήταν τρόπος αυτός να κάνουμε πιο γρήγορα την δουλειά μας. Αν είχαμε το έγγραφο νωρίτερα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός. Οι διαδικασίες πρέπει να πάνε πιο γρήγορα. Πρέπει να προσδιορίσουμε τις διαδικασίες και να τις επιτυχουμε. Για να δούμε λοιπόν, παρακαλώ, η κυρία από την Επιτροπή πρώτα. Ευχαριστώ πολύ σε σχέση με τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητε αυτές για να καταρτιστούν οι, οι, οι απολογισμοί. Οι πληροφορίες σε σχέση με τις αιτήσει καλλιέργειες για τη γεωργία φτάνουν στις 15 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν, να αναλύσουμε τις πληροφορίες αυτές για να καταρτήσουμε μετά τους ε, λογαριασμούς από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κομμάτι που με αφορά και μετά να τους ενοποιήσω με τα διάφορα άλλα όργανα και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Επομένως η διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εικόνα για προσωρινούς λογαριασμούς, απολογισμούς μέχρι τα τέλη Μαρτίου είναι ήδη πολύ πιεστική. Άντε να πω μια εβδομάδα πιο νωρίς, πότε πότε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ε, καταθέτω πιο νωρίς, γιατί χρειάζομαι όλες αυτές τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Και αν δεν φτάσουν, δεν μπορώ να κλείσω την εικόνα από πλευρά τη Επιτροπή για του λογαριασμού. Βέβαια, μπορώ να πω ότι άπαξ και έρθουν στα χέρια μα όλοι οι λογαριασμοί, και βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύει ο καθένα στη δουλειά του, στη γωνιά του. Συνεργαζόμαστε στενά και με του δημοσιονομικού ελεγκτέ και μπορεί να αρχίσει ήδη η δουλειά του δημοσιονομικού ελέγχου. Τα στοιχεία δηλαδή που έχουμε και είναι χρήσιμα για το δημοσιονομικό έλεγχο πηγαίνουν πολύ γρήγορα στο ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά είπα, χωρί τι πληροφορίε των κρατών μελών που είναι απολύτω απαραίτητα, δεν μπορώ να κάνω ε, ούτε για την Επιτροπή τον απολογισμό, ούτε ε, τον ενω, τους ενοποιημένους Και βεβαίως Πρέπει να γίνει και δουλειά σε σχέση με τις λοιπές εκθέσεις επιδόσεων κυρίως και πάλι πρόκειται για πληροφορίες που λαμβάνουμε στο ίδια χρονική περίοδο που πρέπει να δούμε, να συλλέξουμε τα στοιχεία, να τα αναλύσουμε, να τα ενοποιήσουμε, να τα, να τα μετατρέψουμε σε ε, λογαριασμούς που θα εγκρίνει στη συνέχεια η Επιτροπή. Για τους προσωρινούς, προσωρινούς λογαριασμούς είναι πολύ δύσκολο μια προσπάθεια σοβαρή όπως κάναμε και πέρσι θα ήταν να καταθέσουμε νωρίτερα κατά ένα μήνα τον τελικό απολογισμό όπως κάνουμε και φέτος. Δηλαδή τρέχουμε για να προλάβουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουν εγκριθεί τα πάντα. Η μάλιστα. Ναι, όμως μια ερώτηση ακόμα. Με απασχολεί οι εκθέσει αιτήσεων δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το νωρίτερο πότε μπορούν να κατεθούν. 30 Ιουνίου λέει ο δημοσιονομικός κανονισμό, αλλά προφανώς είναι αργά. Εσείς μας λέτε μπορούσατε 30 Μαρτίου να έχετε τις δικές σας. Αλλά αυτές οι εκθέσεις των ε, ειδικές εκθέσεις των γενικών διευθύνσεων το ταχύτερο πότε μπορούν να κατεθούν. Το ενωρίτερο. Γιατί αυτό μας ε, διευκολύνει πολύ εδώ στη δουλειά μας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Το νωρίτερο λοιπόν πότε. Οι αιτήσει εκθέσεις υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουνίου και συνοδεύεται από την έκθεση της ετήσιας απόδοσης και διαχείρισης. Και αυτή την έκθεση εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μια σύνθεση των ετήσιων ε, εκθέσεων δράσεων. Οπότε όλο το πακέτο είναι διαθέσιμο 15 ε, Ιουνίου. Δύο εβδομάδες ε, δηλαδή. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κέρδος θεωρώ χρονικά. Το θέμα είναι Αυτές οι εκθέσεις ε, πότε μπορούν να μας ε, δεδεθούν. Το πότε θα παρουσιαστούν είναι άλλο θέμα. Όπως είπα όμως τα έγγραφα τα οποία εγκρίνουν αυτές τις εκθέσεις όλες είναι η ετήσια έκθεση διαχείρισης και απόδοσης και αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον εγκριθούν όλα τα υπόλοιπα ως πακέτο και είπαμε το αργότερο 15 Ιουνίου και μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα ε, διαθέσει ε, και να, τα, ε, και να δώσει την πρόσβαση στο κοινό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρέκορο. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο και να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τις πληροφορίες ε, που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία του MPR μέχρι τις 15 Ιουνίου και την υποβολή μέχρι τέλη Ιουνίου. Το είχαμε συζητήσει αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είχαμε αναφέρει και σε κάποιες επιστολές που ανταλλάξαμε και νομίζω ότι αυτό προφανώς βοηθάει. Θα μας βοηθήσει σαφώς να ολοκληρώσουμε την ετήσια έκθεση μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Και ίσως καλά θα ήταν να παρουσιάσουμε και τις εσωτερικές μας καταληκτικές ημερομηνίες για την ετήσια έκθεση του 2017 μέχρι τέλη Μαΐου. Υποθέτουμε ότι όλα τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης θα έχουν εγκριθεί και μετά μεταξύ 13 Ιουνίου και 2 Ιουλίου θα έχουμε ε, ένα περιθώριο για τις ιστορικές μας διαδικασίες και υποθέτουμε ότι η τελική έγκριση θα γίνει 12 Ιουλίου. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι έτοιμα τα κεφάλαια να πάνε στη μετάφραση. Μετά έχουμε την ιστορική μας ημερομηνία προθεσμία για να προετοιμαστούν οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές. 31 Αυγούστου είναι αυτή η προθεσμία και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου θα προετοιμάσουμε το τελικό layout και θα γίνει και η τελική επιμέλεια του κειμένου και θα προετοιμαστεί για δημοσίευση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το 2017, την έκθεση του 2017. Και φυσικά, αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε ομάδα εργασία για να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων, με χαρά θα συμμετάσχουμε. Ευχαριστούμε. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και σημαντικό θα ήταν αν είναι έτοιμη η έκθεση στις 12 Ιουλίου. Ανακύπτει το ερώτημα το εξή. Εντάξει, δεν λέω να γίνει διορθώσει, να είναι όλα καλά και έτοιμα. Και μόνο όταν είναι έτοιμη έκθεση θέλουμε να την ε, δούμε, γιατί είναι η πιο σημαντική δουλειά του Ελεκτικού Συνεδρίου αυτή. Αλλά μήπως ε, θα μπορούσε να γίνει δημοσίευση σε μία γλώσσα στην αρχή και μετά να γίνει η μετάφραση και η δημοσίευση και σε άλλες ε, γλώσσες. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει δημοσίευση 12 Ιουλίου σε μία γλώσσα και μετά να ακολουθήσουν οι γλωσσικές για άλλες γλωσσικές εκδοχές. Κοιτάξτε, πιστεύω αυτή η απόφαση θα ήταν στρατηγικής φύσεως και ο πρόεδρος θα έπρεπε να διαβουλευτεί με όλα τα μέλη του σώματος. Όπως είπατε, αυτό ενδεχομένω να χρειαστεί να διαρρήξουμε κάποια ταμπού. Στις εκθέσεις μας συστήνουμε λογοδοσία και μεγαλύτερη λογοδοσία και μιας και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, σύντομα 27, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, ταυτόχρονη παροχή των πληροφοριών αυτών σε όλους. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θα το συζητήσουμε φυσικά με τον Πρόεδρο ιστορικά και ελπίζω να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ναι, αν χρειάζονταν ε, διορθώσεις ή ε, μόνο περιορισμένες ε, διορθώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στο παρελθόν, να προσθέτουμε διορθωτικά σημειώματα για να είναι σωστέ αυτές οι πληροφορίες. Αυτό το δίνω στροφή για σκέψη, γιατί ιδάλω δεν βλέπω πώς θα προχωρήσουμε στην όλη αυτή η ιστορία. Είναι. Ευχαριστώ πολύ. Όντω. υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι ε, έχουν λόγο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής και υπάρχει και ο ρόλος των κρατών μελών ή διάφορες φάσεις της διαδικασίας απαλλαγής. Οπότε Καμιά φορά εμείς, επειδή είμαστε ευρωβουλευτέ, είναι δύσκολο να δούμε την ευρύτερη εικόνα, γιατί εμπλέκονται τόσοι πολλοί οργανισμοί και είναι εύκολο να πει ο ένας, ε, το ένα θεσμικό όργανο, ναι, ας επιταχύνουμε, αλλά εξαρτάται και από τους ρυθμούς των υπολείπων. Ίσως είναι χρήσιμο λοιπόν για μας να λάβουμε κάποιο είδους διάγραμμα που θα παρουσιάζει ε, τα στάδια της διαδικασίας ε, απαλλαγής ε, και όπου θα αναφέρεται ποιος είναι υπεύθυνο για κάθε φάση για να δούμε πού υπάρχουν ευκαιρίες επιτάχυνσης και ποιος θα μπορούσε να κάνει τι. Ίσως η γραμματεία θα μπορούσε να το αναλάβει σε αυτή τη φάση. Οπότε αν δούμε ολόκληρη την εικόνα, ίσως θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε πού υπάρχουν δυνατότητες επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας. Μάλιστα, το σημειώνουμε. Η κυρία Γέλα Άκουσα τη συζήτηση και νομίζω πως υπάρχει μια σειρά πληροφοριών που καμιά φορά ε, λαμβάνουμε δύο και τρεις φορές ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και καταλαβαίνω πως χρειάζεται να εξορθολογήσουμε και να απλοποιήσουμε τα ερωτηματολόγια. Το κάναμε για τους εξωτερικούς οργανισμούς και είδα πως ε, φέτος ο εισηγητής, ο κύριος Σαρβαμά, ε, έθεσε εκ νέου το θέμα αυτό. Πιστεύω λοιπόν πως ε, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, ένα βασικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα συμφωνήσουμε για το ποιες είναι οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες και σε σχέση με ποιο έτος διανύουμε, να κάνουμε και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, είτε για τα συγκεκριμένα θέματα που τρέχουν εκείνο τον χρόνο, είτε για κάτι το οποίο θα προκύψει ε, τη χρονιά εκείνη ή κάποιες επόμενες. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, γιατί ε, νομίζω ότι η κρίσιμη στιγμή είναι ο Ιούνιος. Και ίσως θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε και κάποιες από τις δικές μας ακροάσεις, για παράδειγμα, έτσι ώστε όλη η διαδικασία να κλείνει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης, ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε, έτσι ώστε το ερωτηματολόγιο να γνωρίζουν οι εξωτερικοί οργανισμοί πως ε, θα καλύπτει κάποια στοιχεία κλειδιά και μετά θα πρέπει να συμπληρώνουν και με επιπλέον στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, και θα ήταν πολύ θετικό αυτό, γιατί θα ήταν και ένα είδους πίεση για να βελτιωθούν οι διαδικασίες, παράδειγμα για τις πληροφορίες που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο θα βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές πιο γρήγορα και επίσης θα βοηθούσε και το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί εδώ βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο που έχουμε τη μεθοδολογία την παραδοσιακή και τη μεθοδολογία της παρουσίασης ε, των ενοποιημένων λογαριασμών, για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Μπορούμε να το συζητήσουμε και με τους συντονιστές, το κάνω εδώ στην ομάδα και να δούμε αν θα μπορούσε ε, παράλληλα να τρέχει φέτος εκτός από την απαλλαγή και μία ομάδα εργασίας με τους θεσμούς με τους οποίους είναι απαραίτητο να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και επαναλαμβάνω να τρέχει παράλληλα με την απαλλαγή φέτος και να δούμε τα βασικά στοιχεία, όχι να συγγράψουμε ένα τεύχος ε, ως νέα βίβλο για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο ελέγχου και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποια σημεία μπορούμε να επιταχύνουμε, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες και έχουμε και πληροφορίες που λαμβάνουμε και στοιχεία του πρώτου εξάμεινο Και που δεν χρειαζόμαστε πολύ. Και όταν έχουμε το έγγραφο του follow-up για την προηγούμενη απολογή, μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και άλλες φορές ήδη ε, βρίσκονται αυτό στην έκθεση για την διαχείριση και την απόδοση του τρέχοντος έτους. Οπότε, ας μην περιμένουμε εμείς τόσο πολύ όταν το follow-up φτάνει καθυστερημένα. Έτσι ώστε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να έχουμε κάνει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς έτσι ώστε για το δεύτερο εξάμεινο να έχουμε μόνο αυτό που είπατε κι εσείς. Ε, σφάλματα τα οποία εντοπίζονται, διορθώνονται, προσθήκες και αν, ε, ε, αν δημιουργηθεί η ομάδα εργασίας βεβαίως και οι σκιώδες θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Πώς σας φαίνεται. Η πρόθεσή μου ανεξάρτητα από το θέμα του χρονοδιαγράμματος ήταν να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πιο απλή διαδικασία, χωρίς βεβαίως η διαδικασία αυτή να είναι λιγότερο απαιτητική. Γιατί έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και πολλές φορές ζητάμε ακόμα περισσότερες και έχουμε επικαλύψεις παρόλο που γνωρίζουμε είτε μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε ακόμα και από τους ίδιους εξωτερικούς οργανισμούς, πως τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα, παρόλο που δεν έχουν πάρει τη σφραγίδα την τελική, ας πούμε. Αν λοιπόν το επιθυμείτε κι εσείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να ευχαριστήσουμε και το Ελληνικό συνέδριο για την καλή του διάθεση. Και να γίνεται παράλληλα αυτός ο διάλογος και η προσπάθεια επιτάχυνσης. Νομίζω ότι αν το αποτύχουμε αυτό στο επόμενο έτο, στο νησιν ε, θα πρέπει να δούμε από την αρχή πώ θα προσαρμόσουμε την διαδικασία. Πώ μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε την καλλιτική ημερομηνία και ανάλογα όλε τι προηγούμενε ε, προθεσμίε. Ε. Και αυτό προφανώ εξετάζεται και το Συμβούλιο και από πολλού άλλου παράγοντε του οποίες δεν θα πρέπει να του υποτιμούμε. Ε, αλλά εμεί τουλάχιστον μια πρόταση πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το δικό μας τμήμα. Γιατί ω τώρα η διαδικασία χωρίς απαλλαγής ήταν το Μάη. Τώρα το πήγαμε Μάρτιο. Ελπίζω σιγά σιγά να φτάσουμε στον Ισηνένα. Να κάνουμε μία πρόταση. Τώρα, το θέμα της τυποποίησης ε, των ερωτηματολογίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα άλλα θεσμικά όργανα. κοιτώντα τι προβλήματα διαφορετικά και τι ξεχωριστά χαρακτηριστικά έχουν οι διάφορες υπηρεσίες, τα ταμεία. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πραγματική τυποποίηση στις εξωτερικές υπηρεσίες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά προς το συμφέρον μας είναι. Και γι' αυτό λοιπόν στην τελευταία αναθεώρηση ε, της διαδικασίας χωρίς απαλλαγές, είπαμε ότι κοιτάξτε αυτές τις πληροφορίες τις χρειαζόμαστε στάνταρ κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να τις να θέτουμε σχετικά αιτήματα κάθε φορά για να υπάρχει σαφήνεια και έχω δύο κακές ειδήσει και μία καλή για την Επιτροπή. Μία κακή ειδήση είναι είμαστε η Επιτροπή με τις πιο πολλές συνεδριάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερον, ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλαγή προϋποθέτει Ανάγνωση 8 μέχρι 9.000 σελίδων. Φυσικά δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όποιος προσπαθήσει να κατακτήσει αυτές τις 9.000 ε, ε, σελίδες και τώρα έχετε η καλή είδηση, πραγματικά ξέρει τι συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε ταμείο, σε κάθε θεσμικό όργανο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχετε υπόψη, να ξέρετε τι, τι γίνεται και τι λένε κάποια βασικά έγγραφα για τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Και αν αυτές οι εκθέσεις δημοσιεύονται πιο νωρίς, έστω και ανεπίσημα, το Μάρτιο για παράδειγμα, μέχρι τέλη Μαρτίου, αλλά τελικά καταλήγουν στο συρτάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι 15 Ιουνίου για ιστορικούς λόγους. Δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας. Θα πρέπει να τις έχουμε τις ε, πληροφορίες αυτές νωρίτερα στη διάθεσή μας, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα αυτά έργα. Και αν αυξηθεί και η έρευνα, αν έχουμε και το θέμα της ΔΕΦΚΟ, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει πολλά. Η Γενική Διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε σίγουρα να είναι καλύτερη, γιατί κάθε χρονιά μου λείπουν πληροφορίες και εκνευρίζομαι. Είναι σημαντικές αυτές λοιπόν οι πληροφορίες και η διστάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λογοδουσία ή όχι. Το θέμα που έθιξε η κυρία Αγιάλα Σέντερ, ε, το θέμα της ομάδας εργασίας, είναι σημαντικό να υπάρξει ομάδα εργασίας. Γιατί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας. Να δούμε μήπως ε, καλό θα κάναμε να καλέσουμε την Προεδρία και να θέσουμε και ένα γραπτό ερώτημα. Μια, μια γραπτή ερώτηση προς την ε, Προεδρία και να δούμε τι έχει να μας πει. Το θέμα των εξωτερικών υπηρεσιών, το θέμα του ελεκτικού συνεδρίου τώρα. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε και ότι θα πρέπει τη δικασία να καταρτιστεί εκ νέου από την αρχή θα πρέπει ενδεχομένω ε, να γίνει ακρόαση διάφορων επιτρόπων σε μία συνεδρίαση. Έτσι πως είναι τα πράγματα όμως δεν ε, γίνεται. Ενδεχομένως ε, να προηγηθούν οι εξωτερικές υπηρεσίες για να έχει πιο μεγάλο περιθώριο κάπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε διάφορα μοντέλα. Αλλά μετά, με τι προθεσμίε που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. είναι Έχετε δίκιο και για το πόσο πολλή δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι συχνά βλέπουμε πως είναι οι ίδιες πληροφορίες αλλά σε διαφορετικές εκθέσεις. Οπότε καλό θα ήταν να εξορθολογήσουμε στο μέγιστο δυνατόν, έτσι ώστε αν είναι να διαβάσουμε 8.000 σελίδες, να είναι 8.000 σελίδες με διαφορετικά στοιχεία, όχι τα ίδια σε άλλα κεφάλαια, γιατί πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η έκθεση του follow-up έχει μεγάλη ε, ταύτιση με την έκθεση για την απόδοση της προηγούμενης χρονιάς και στα ερωτηματολόγια ξαναρωτάμε στοιχεία τα οποία ήδη έχουμε. Οπότε καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια των υπολείπων οργάνων και των ε, μελών μας να δούμε τι δεν χρειαζόμαστε. Γιατί αν οι 8.000 μπορούν να γίνουν 3.000, γιατί απλώς οι 8.000 τα βλέπουν από διαφορετική οπτική γωνία, καλό θα ήταν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί έτσι, χωρίς να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Γιατί αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει πολλές φορές, παρόλο που υποβάλλουμε πολλά αιτήματα, ε, να λάβουμε την πληροφορία που θα μας εξηγήσει ε, κάποια απορία. Αυτά τα λέω γιατί σκοπός μας είναι να εξορθολογήσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε. Ähm, ναι, βεβαίω και είναι απολύτως απαραίτητο για όλους και όλοι γνωρίζουμε ότι του χρόνου οι συνάδελφοι θα ασχολούνται επιτοπλίστων με άλλα θέματα. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και πάνω απ' όλα και στο θέμα της ε, τυποποίησης των εργασιών. Μπορούμε μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχουμε έγγραφα που είναι πολύ σημαντικά για μας, αλλά για να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε πρέπει να έχουμε πρόσβαση και σε πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ξέραμε από την αρχή ότι δεν ήταν παιχνιδάκι και βόλτα στο πάρκο έλεγχος του προπολογισμού. Το κλείσαμε το θέμα αυτό. Στη ημερήσιας δέταξη. σας ευχαριστώ αν δεν θέλετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ τους παρόντες και βεβαίως ξέρω ότι τους... Ε, είναι, ιδιαίτερο μέλημα και για εκείνους η βελτίωση των διαδικασιών, η συντόμευση των χρόνων. Ευχαριστώ πολύ και έτσι πάω στο σημείο 9. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ είσαστε. Α, ωραία, δεν κολλήσατε λοιπόν στην κίνηση. Μπράβο, που είσαστε όμως. Α, εντάξει. Οκ. Okay. Κύριος Βαλέριο Μπλάκο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για την παρακολούθηση της επαλλαγής του 2016. Και δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Μπλάκο να μας περιγράψει συνοπτικά την κατάσταση, πώς το βλέπετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκλήθημε να, συζητήσουμε μαζί σας τις συνέπειες της απόφασης ε, του δικαστηρίου του Ιανουαρίου του 2018 αποφάσεως με την οποία ανέρεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απόφαση του δεύτερου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου Δημοσίας Διοικήσεως για μία σύνθεση με συμμετοχή του δικαστού Αλεξάνδερ Κόρνεζοφ, του οποίου ο διορισμός είχε θεωρηθεί ως πλήμελης για λόγους τυπικούς, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διαπιστώσει ακυρότητα της σύνθεσης, της απόφασης μάλλον, του ε, Γενικού Δικαστηρίου λόγω μη σύνθεσης. Και αυτό το βλέπουμε να αντικατοπτρίσετε στο σημείο 53 της απόφασης για την απαλλαγή όπου καλείται να προσδιορίσει ποια απόφαση του δεύτερου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου Δημοσίας Διοίκησης με την επίμαχη σύνθεση επηρεάζεται από αυτή την απόφαση του Μάλλον ποιες είναι οι αποφάσεις στον πληθυντικό που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι δικαιοδοτικές αποφάσεις ισχύουν μέχρι ότου αναιρεθούν ή ακυρωθούν από το ανώτατο δικαστήριο, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προς το παρόν μόνο η εν λόγω απόφαση έχει ακυρωθεί, η εν λόγω απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Μόνο αυτή δηλαδή αφορά η διαπίστωση μη νόμιμη σύνθεση του δικαστικού σχηματισμού από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, εκκρεμούν αρκετές ε, αιτήσεις αναιρέσεως, 8 μέχρι τώρα, σχετικές με αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, εκ των οποίων δύο μόνο αφορούν σύνθεση του Γενικού Δικαστηρίου Δημοσίας Διοικήσεως με συμμετοχή του ίδιου δικαστού, εκείνου δηλαδή του οποίου το διορισμό ε, συζητεί η απόφαση αυτή του Ιανουαρίου του 2018. Επομένως, αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, δύο ακόμη αποφάσεις του, δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μπορούν, μπορεί να αναιρεθούν, ενδέχεται να αναιρεθούν, με βάση τους ίδιους λόγους. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες αποφάσεις και διαταγές που έχει υπογράψει ο ίδιος δικαστής, χωρίς όμως να έχουν προσβληθεί με αίτηση ε, αναιρέσεως και τώρα πια καλύπτονται από το δαδικασμένο και εκ τούτου δεν μπορούν να ε, προσβληθούν. Μια πρώτη απάντηση λοιπόν είναι αυτή ως απάντηση στο σημείο 13 του ψηφίσματος για την απαλλαγή. Αλλά βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το θέμα. Αυτό είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Είσαστε υπεύθυνος για διοικητικά θέματα στο δικαστήριο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είχαμε αυτά τα θέματα να συζητήσουμε. Είναι καλό να γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι πρόκειται και η υπόθεση είναι ότι υπήρξε μια απόφαση που προσβλέπει που προσβλήθηκε επειδή είχε γίνει διορισμός δικαστή τέσσερις μήνες πριν από την ολοκληρώση της διαδικασίας και εδώ είπε ξεκάθαρα με την απόφαση για ανέρεση στο δικαστήριο ήταν παράνομος ο διορισμός του δικαστή επομένως κρίνει μη νόμιμη τη σύνθεση του δικαστικού σχηματισμού εδώ είναι και το Συμβούλιο το οποίο είχε κάνει το διορισμό και διαπιστώνει το δικαστήριο ότι κάθε απόφαση στην οποία έχει συμμετάσχει ο δικαστή αυτής αυτός είναι παράνομη. Από ό,τι καταλαβαίνω, από τις έξι αποφάσεις οι τέσσερις μας λέτε έχουν προσβληθεί. Ε, το γεγονός ότι γίνεται ένας διορισμό μέσα στο τετράμινο πριν από την ολοκλήρωση μια διαδικασία και βέβαια αυτό έχει και το κόστος του, δείχνει πόσο κακά λειτουργούν οι διαδικασίες. Δεν ε, μπορώ να διανοηθώ ότι οι νομικοί δεν αντελήφθησαν ότι μια τέτοια μορφή διορισμού μέσα από ένα κατάλογο υποψηφίων του 2013 που είχε εκδοθεί για να καλυφθούν θέσεις άλλων δικαστών που αποχωρούσαν ε, μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη. Δεν θα έπρεπε οι νομικοί από εσά να έχουν επισημάνει στο Συμβούλιο ότι δεν είναι ο διορισμός αυτός νόμιμος όπως τα όφυλα. Έχετε κάτι να απαντήσετε. Και για όλα αυτά τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με, τον, ε, με το έργο του Βούλγαρου δικαστή, δηλαδή με, με τις συνέπειες που μπορεί να έχει παρουσία του Βούλγαρου δικαστή σε άλλες εργασίες. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν ε, ε, πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να παρεμβαίνει στον ορισμό των μελών του, που είναι αρμοδιότητα άλλου θεσμικού οργάνου, εν προκειμένου του Συμβουλίου. Επιπλέον, το δικαστήριο δεν μπορεί να προδικάσει ζητήματα νομικά που μπορεί εκ των υστέρων να προκύψουν. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υποχρεούμε σήμερα να περιοριστώ ε, στα όσα μπορώ να σας πω, διότι ως εκπρόσωπος του δικαστηρίου μπορώ να σας δώσω κάποια πραγματολογικά στοιχεία. Αλλά νομική ανάλυση, όχι. Γιατί μπορεί πάντα να είναι κάτι τέτοιο αντικείμενο προσφυγής ή ε, έτσι συναρέσεως ενώπιον του δικαστηρίου. Στο συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπρεπε να το διευκρινίσω. Στα αριθμητικά στοιχεία που σας έδωσα νωρίτερα, καθώς δεν πρόκειται για τέσσερις υποθέσεις και παραλαμβάνω σύνθεση δικαστική του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με συμμετοχή μεταξύ των δικαστών του κυρίου Καρνεζόφ ήταν 21 τον αριθμό οι αποφάσεις στις οποίες συμμετείχε ο κύριος Καρνεζόφ. Πέρα της ανερεθήσας απόφασης όμως μόνο δύο έχουν ανερεσιβληθεί και άρα συνολικά Μπορούμε να έχουμε μόνο τρεις εν όλο αποφάσεις που μπορεί να αναιρεθούν. Άρα είναι μάλλον ολίγες. Καλώ ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Είπα, ε, αυτό είχα σημειώσει και εγώ. Δύο προσφυγές και δύο ετήσεις αναιρέσεως. Καλά, ευχαριστώ για τη διόρθωση και τη ευκρίνηση. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε ένα δικαστή τώρα, ο οποίος παραμένει όμως στο δικαστήριο. Έχει γίνει μια προκήρυξη η οποία βεβαίως απαιτεί και πείρα, επαγγελματική. Ο δικαστής από τη Βουλγαρία λοιπόν κάνει αίτηση επικαλούμενος την ε, επαγγελματική του πείρα και είχε ένα πλεονέκτημα για την ανάληψη ε, καθηκόντων στο ίδιο το δικαστήριο, πλεονέκτημα που είναι η επαγγελματική αυτή πήρα σε ένα εργατοδικείο, το οποίο πλεονέκτημα δεν προσέφερε κάποιος άλλος υποψήφιος από τη Βουλγαρία. Τώρα με την απώλεια αυτής της δυνατότητας ή μάλλον η, επιλογή αυτού του δικαστού σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε από το γεγονός ότι διέθετε αυτή την επαγγελματική πείρα από το εργατοδικείο. Πρόεδρε, το δικαστήριο επανέρχομαι και θα το ξαναπώ. Δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία διορισμού του κυρίου Κορενζόφ ως δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο Δημοσίας Διοίκησης. Ο διορισμός έχει να κάνει με τα άρθρα 254-255 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτά απορρέει ο διορισμός από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι οποίες υιοθετούν την απόφαση με βάση την υποψηφιότητα που προτείνει το ε, οικείο κράτος μέλος και δεν έχει τίποτε να πει το δικαστήριο ε, εκ τούτου δεν μπορεί να πει καθόλου ε, ενώπιον σα το πόσο αυτή η τετράμινη εμπειρία επηρέασε ή όχι το διορισμό. Δεν με ξαφνιάζει πρέπει να πω η απάντησή σας, αλλά επιτρέψτε μου να, επι, να επιμείνω. Γιατί αυτό έχει ζητήματα. Και ρωτώ, εγώ σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για να καταλάβω αυτή η δουλειά στο ε, εργατοδικείο σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει την επιλογή. Υπάρχει κάποια ομάδα, κάποια επιτροπή, ποιος ήταν ο πρόεδρος, σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει αυτή η επαγγελματική πείρα. Γιατί εν τέλει ξέρετε πιο από όλα αυτά σημασία έχει το αν έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες από την επαγγελματική αυτή πείρα ή όχι ο ε, δικαστής από τη Βουλγαρία. Απάντηση. Ο διορισμός ε, δικαστή ως διαδικασία είναι κάπως διαφορετική ε, με την εξή έννοια. Δεν έχουμε μια πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητων σαν αυτή που αναγράφεται στη συνθήκη. Οπότε όταν μιλάμε για διορισμό ε, στην περίπτωση του δικαστή από τη Βουλγαρία δεν είναι απαραίτητο όπως είχαμε και άλλες υποψηφιότητες οι οποίες θα είχαν ληφθεί υπόψη στα πλαίσια μιας επίσημης διαδικασίας. Πρόκειται για εσωτερική διαδικασία του κράτους μέλους ε, και δεν γνωρίζω ακριβώς πώς έγινε. Ίσως θα μπορούσαμε ε, στην Επιτροπή άρθρο 255 να υποβάλουμε το εξής ερώτημα γιατί εκεί μίλησε η Επιτροπή αυτή για την ισοδυναμία της υποψηφιότητας Κορνιζόφ και για το κατά πόσο ε, μπορεί να διοριστεί ε, στο δικαστήριο. Εγώ δεν μπορώ να υποκαταστήσω την Επιτροπή αυτή και δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση για το κατά πόσο αυτή η τετράμινη εμπειρία λήφθη υπόψη και με ποιο τρόπο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ποιον θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε λοιπόν. Ε, για μια φορά ακόμα, η διαδικασία διορισμού ε, περνάει από τη φάση του ορισμού υποψηφίου από το κράτος μέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να απευθυνθείτε στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον επικεφαλής ε, της ε, Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων. Μιλάτε πάντα για την Επιτροπή Άστρου 255. Νομίζω την Προεδρία την τελευταία φορά την είχε, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά θα, θα, σας, το, θα σας ενημερώσω. Ο κύριος Μάρκ πώς ήταν νέο, ναι, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος. Ναι. Ναι. Χαίρομαι λοιπόν που το διευκρινίσαμε και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Ξέρετε, είναι περίεργο ότι έχουμε διαδικασίες για εκλογή των δικαστών που προφανώς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και διαπιστώνουμε ότι υπονομεύονται οι διαδικασίες αυτές. Οι διαδικασίες αυτές. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, συμπτώσεις ε, στη ζωή και στην πολιτική και στο θέμα αυτό της ε, παρανομίας ε, και το πόσο ακολουθήθηκε η διαδικασία για την εκλογή δικαστών. Φυσικά δεν μιλάμε για, τετράμινη, για μια τετράμινη για διορισμό. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται στο μέλλον και τι διαδικασίες θα τηρηθούν στο μέλλον. Και είναι κρίμα που το δικαστήριο λέει, ε, τι να κάνουμε, να τα σβήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή το δικαστήριο δεν νοιάζεται, δεν το ενδιαφέρει η διαδικασία αυτή. Εμείς πώς θα το εκλάβουμε αυτό. Κυρία Πρόεδρε, βεβαίω όλοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό και στο δικαστήριο και εκτός, αλλά μην ξεχνάτε πως δεν έχει το 10 καμία αρμοδιότητα σε επίπεδο ορισμού των μελών του. Και γι' αυτό υπογραμμίζω πως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά καθόλου την απαλλαγή. Παρόλο που έχει τοποθετηθεί το σημείο αυτό στην απόφαση, στο ψήφισμα απαλλαγή, μπορώ να σας δώσω πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μα και μπορώ να σα δώσω και πληροφορίε για την απόφαση που έχει εκδοθεί, αλλά το διορισμό αυτό δεν τον αποφάσισε το δικαστήριο και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Εσείς απευθύνεστε στο δικαστήριο, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το θέμα. Στην παρούσα φάση δεν έχω κάποιον ε, στόχο, ε, δεν έχω κάποιον στον επίκεντρο της προσοχής μου, αλλά κάνω ερωτήσεις. Ε, γιατί αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει περάσει χωρίς να δώσουμε προσοχή και δεν έχει τεθεί το θέμα αυτό. Δεδομένων συνθήκων τις οποίες θεωρώ πολύ αμφίβολες. Το θέμα λοιπόν της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας τίθεται. Φυσικά είμαστε υπεύθυνοι για τις ε, οικονομικές συνέπειες των δράσεων και εδώ μπορούμε να αποδείξουμε ότι και υπήρξαν οικονομικές συνέπειες και ενδεχομένως να υπάρξουν περαιτέρω οικονομικές συνέπειες. Προέκυψε πολύ σημαντικό κόστος και για το φρολογούμενο χωρίς να υπήρχε οποιοδήποτε λόγος, οποιαδήποτε αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την απόφαση αυτή, σε ό,τι αφορά και τις μερωτικές αποφάσεις θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κυρία Πλάκα που ήλθατε στην Επιτροπή μας και πολύ φοβάμαι ότι θα παραμείνουμε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε στο σημείο 8. Την ειδική έκθεση 10-2008 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς. Η κυρία Κλάουτα Σμίτ είναι η εισηγήτρια και ο κύριος Ζωάο Φιγκερέιδο είναι ο αρμόδιος ε, από το Ελληνικό Συνέδριο και έχουμε φυσικά και τους ε, ε, συναδέλφους ε, από την Επιτροπή Άγκρη μαζί μας. Κύριε Βιγγερέρο, αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τιμή μου. It's an honor. Thank you. Thank you. It's an honor and also a pleasure. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας δώσω μία απαντική απάντηση στο αίτημα σας για την παρουσίαση της ε, έκθεσης ελέγχου μετά την ε, συντομότερη παρουσίαση που έκανα πριν από κάποιες εβδομάδες. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση σε PowerPoint και σας παρουσιάζω τα τελικά απορίσματα και τις συστάσεις προς την Επιτροπή για το βασικό καθεστώς ενίσχυσης ε, για τους γεωργούς. Θα σας παρουσιάσω κάποιες γενικές, ε, γενικά συμπεράσματα και να σας πω καταρχάς ε, ότι το καθεστώς βασικής ενίσχυσης του γεωργούς είναι σε καλό δρόμο. αλλά έχει περιορισμένη συμβολή σε ό,τι αφορά την απλούστευση τη στόχευσης για τη σύγκληση των επιπέδων ενίσχυση σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των ε, επιδοτήσεων. Καταλήξαμε στα εξή συμπεράσματα. Οι υπηρεσίε παροχή πληρωμών κάνουν σημαντικέ προσπάθειε για να δρομολογήσουν το νέο αυτό σύστημα που προέκυψε από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Τα συστήματα ελέγχου στα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε ε, μετρίασαν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και εκχωρήσεων τέτοιων ε, επιδοτήσεων. Οι πληρωμές BPS ε, δεν επηρεάζονται σημαντικά από σφάλματα, όπως αναφέρουμε και στην ετήσια έκθεση για τα αίτια αυτά. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι τιμές BPS ήταν ανακριβείς ήταν προσωρινός υπολογισμός τους ε, βάσει κάποιων εκτιμήσεων και κάποιες υπηρεσίες ε, παροχής πληρωμών αντιμετώπισαν δυσκολίες. Να δούμε λοιπόν γιατί. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του νέου αυτού συστήματος ε, βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς, διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εκτενή καθοδήγηση προς τα κράτη-μέλη. Και οι έλεγχοι είχαν καλά αποτελέσματα αλλά πιστεύουμε ότι έλειπαν κάποιες ε, πληροφορίες σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει ζητήσει πιο πολλά από τα όργανα πιστοποίησης, από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, το σκέλος της απλούστευσης, να σας υπενθυμίσω ότι η απλούστευση ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης αλλά οι ευρωπαϊκοί κανόνες περιλαμβάνουν πολλές ε, δυνατότητες και εξαιρεσει. και σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη δεν επέλεξαν την οδό της απλούστευσης. Βλέπετε ένα παράδειγμα εδώ. για ένα κράτος μέλο και τις επιλογές που έκανα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των γεωργικών εκτάσεων. Σε διάφορους τομείς ε, ε, υπήρχε αλληλεπικάλυψη διάφορων γεωργικών περιφερειών. Και επίσης αυτές οι πολλαπλές δυνατότητες επέτρεψαν ε, μεγάλο κέρδος για κάποιους γεωργούς σε ό,τι αφορά τη στόχευση τώρα. Ένα στόχος τη μεταρρύθμισης ήταν αυτό επίση. να υπάρξει καλύτερη στόχευση των ε, γεωργών δημιουργήθηκε ο όρος του ένεργου γεωργό. Σημειώθηκαν κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά γενικά μας δυσκόλεψε και ήταν και περιορισμένος ο αντίκτυπος της πρότασης αυτής. Και γι' αυτό λοιπόν από φέτος τα κρατημέλη, μετά από αποφάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κρατημέλη λοιπόν μπορούν να μειώσουν τα κριτήρια με τα οποία οι ετούντες μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ενεργοί γεωργοί με μια αρνητική λίστα. Σε ό,τι αφορά τη στόχευση, επίσης, ε, διαπιστώσαμε ότι η μεταρρύθμιση ε, επέκτηνε τις κατηγορίες ε, γεών για την παροχή επιδοτήσεων με μια ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα και κάποια κρατημέλη είχαν ενεργή προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου, αλλά οι νέοι κανόνες δημιούργησαν και δυσκολίες ό,τι αφορά την εφαρμογή, πιστεύουμε εμεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύγκληση των επιπέδων ενίσχυσης και τον ε, αυτό αποτέλεσε ασφαλώς βασικό στόχο της μεταρρύθμισης. Με, τα, με τη μεταρρύθμιση ε, τα επίπεδα ενίσχυσης ανά εκτάριο ήταν πιο ενιαία, αλλά τονίζουμε στην έκθεσή μας ότι σε 11 από τα 18 κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές και μετά το 2019. Βλέπετε στο χάρτη τις διάφορες λύσεις και τις διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν το 2019. Η, το καθεστώς βασικής ενίσχυσης έχει περιορισμούς ό,τι αφορά τα θέματα εισοδημάτων που ανησυχούν τους αγρότες και κλείνει και τίνει να προτιμά και να ευνοεί τις μεγαλύτερες καλλιέργειες. Και η απουσία μια βασικής γραμμής και των σαφών στόχων είναι η μεγάλη δυσκολία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της σωστής ενίσχυσης. Και έτσι λοιπόν προτείνουμε προς την, προτείνουμε προς την Επιτροπή τα σε εξής συστάσεις. Καταρχάς, να αντιμετωπίσει τις, αδυναμίε αδυναμίες σε βασικούς ελέγχου, Να βελτιώσει τα... να διορθώσει μάλλον τα δικαιώματα όπου υπάρχει περιθώριο σφάλματο και να αναθεωρήσει συστήματα τα συστήματα για την παροχή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, γιατί είδαμε σκεπτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Επίσης, να βρει λύσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση της υποχρεωτικής παροχής πληροφοριών από τα κράτη-μέλη. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι ρόλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σωμάτων πιστοποίησης σε ό,τι αφορά τα νέα αυτά συστήματα βασικών πληρωμών. Πιστεύουμε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτού κάνει οποιαδήποτε πρόταση για τη μελλοντική σχεδιασμό τη ΚΑΠ, θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση του συστήματο παροχή ενίσχυση σε όλε τι ομάδε γεωργών, να ορίσει του λειτουργικού στόχου για οποιοδήποτε μηχανισμό υποστήριξη εισοδήματο και να εξετάσει πώ μπορεί να πετύχει με τον καλύτερο τρόπο αυτέ του στόχου και να συνδέσει οποιοδήποτε μέτρο σε λειτουργικούς στόχους, με λειτουργικούς στόχους και βασικές τιμές για την σύγκριση της απόδοσης με την οποία θα συνδεθεί η ενίσχυση. Αυτά ήταν τα πιο βασικά πορίσματα κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και οι συστάσεις που θα πρέπει να διαβιβάσουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αποτεχθεί κάποια εξ αυτών ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν έχει εγκρίνει τις συστάσεις που τις έχουμε απευθύνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και περιλαμβάνει και καλύπτει τεράστιο όγκο επιδοτήσεων και δικαιωμάτων. Η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την τόσο διεξοδική ε, έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό όταν δίνουμε τόσα χρήματα να ελέγχουμε και προσεκτικά τη διάθεσή τους. Πρόκειται βέβαια για μια έκθεση που περιμένουμε και μια ειδική έκθεση για την ε, για τις ενισχύσεις στη γεωργία. Θέλουμε να γνωρίζουμε δηλαδή επακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι για τους οποίους ε, δεν, γιατί μάλλον οι στόχοι και η υλοποίησή τους δεν έχουν μετρηθεί, δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν επαρκώς. Ίσως τελικά να φταίει το ότι είναι πολύ μεγάλο η σαν στα κράτη-μέλη ή αλλιώ, και αυτό βέβαια πάντα είναι ένα πρόβλημα για μένα, επειδή επιβαρύνεται υπερβολικά η δημόσια διοίκηση. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει για να δώσουμε το ταχύτερο δυνατό λύσεις. Και από την άλλη βεβαίω βλέπω με ικανοποίηση του γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει βρει τον τρόπο να περιγράψουμε απόλυτη ακρίβεια και περίφραστα την κατάσταση ε, σε σχέση με την γεωργία και την υπεθρογία, τη βασική ενίσχυση. Ε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ο στόχος για την εξασφάλιση αποδοτικής παραγωγής τροφίμων δεν έχει μεταφραστεί σε έναν μετρήσιμο στόχο, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε αν υλοποιείται. Δεν βλέπουμε δηλαδή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ενίσχυσης σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ε, λειτουργίας των επιχειρήσεων ως όρους μετρήσιμους. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι ο επιμερισμός των ενισχύσεων στον πληθυσμό της υπαίθρου, ε, ο επιμερισμός εκείνος ο οποίος θα είναι ο πιο αποδοτικός, ο πιο αποτελεσματικός, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί καλή παραγωγή τροφίμων ε, για τον πολίτη. Και πολλές από τις συστάσεις του συνεδρίου πιστεύω οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε και ότι είναι πολύ ε, υψηλή η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις δημόσιες αρχές πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του δικαστηρίου και να ε, μελετούμε κάθε δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι πολύ διαφορετική βέβαια η εικόνα που παρουσιάζουν τα διάφορα κράτη μέλη. Παραδείγματι για τη Σουηδία πρέπει να μεριμνήσουμε το χέτερο δυνατό ε, ώστε να οριστεί ενιαία το νομικό πλαίσιο για την κατάθεση, για την διάθεση των ε, ενισχύσεων προς τους δικαιούχους παρά είναι μεγάλο το περιθώριο η διακριτική ευχαίρεια δηλαδή που αφήνει το σύστημα στα κράτη-μέλη και οι διαφορετικές επιλογές που έχουν στα χέρια τους ε, οι εθνικές αρχές Οπωσδήποτε θα υποστηρίξω τις συστάσεις υπαριθμών 2 και 3 που είναι πολύ σημαντικές. και επισημαίνουν ε, σε σχέση με τις μελλοντικέ εξελίξεις, κάτω το οποίο βεβαίως ε, ελπίζουμε να μην υλοποιηθεί, αλλά εάν δούμε το 2020 ακόμη περισσότερες περικοπές θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι η ασφάλεια των τροφίμων, η ποιότητα της παραγωγής, η, τα ποιοτικά παραγόμενα τρόφιμα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτός είναι ο ρόλος Γεωργίας και βεβαίως εάν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο ίδιος με τον ε, διαχειριστή πρέπει να γίνεται πολλαπλή καταγραφή και ανάλυση των λογαριασμών, η απόδοση των λογαριασμών αλλά και πάλι παραλαμβάνω χωρίς επιβάρυνση επιπλέον των εθνικών αρχών, γιατί έχουν αρκετή ήδη. Πρέπει να κοιτάξει την εισοδηματική κατάσταση όλων των ιδιοκτητών των γεωργικών επιχειρήσεων, το δυναμικό των εκτάσεων, των διαφορών μεταξύ των εκτάσεων, είτε για, γεωγραφική, είτε για γεωργική συνομιλία παραγωγή, είτε για οικολογική ανάπτυξη, παραγωγή τροφίμων μέσα από την ε, γεωργική δραστηριότητα που οδηγεί σε εισοδήματα, αλλά και άλλα μη γεωργικής προελεύσεως εισοδήματα. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει να επισημάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να κοιτάμε πάντα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, δεν ε, δίνουμε τίποτε ε, δωρεάν. Πρέπει πάντα να κοιτάμε με μεγάλη προσοχή που έχουν δαπανηθεί και με ποιου όρους τα κονδύλια, έτσι ώστε οι ενισχύσεις και αποτέλεσμα να φέρνουν και στοχευμένες να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάτιμπαχ, Ευχαριστώ πολύ καταρχάς το ελεγκτικό συνέδριο για την παρουσίαση αλλά και την κυρία Σμιτ για, την, ε, για τα σχόλιά της που και εγώ υποστηρίζω και υπογραμμίζω στο σύνολό τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις αναλύσεις, τι τις εισοδηματικές αναλύσεις το ταχύτερο δυνατό. Ιδάλλως ε, ε, φαίνεται σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί και να πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς αυτά να στρέφονται προς τους στόχους για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί. Πρέπει να είναι πολύ ε, συγκεκριμένη η επιδίωξη των στόχων και εδώ έχουμε να κάνουμε με 18 δισεκατομμύρια ευρώ που επιμερίζονται σε 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Ε, δεν βλέπω να υλοποιούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις. Το λέει και η κυρία Σμίτα άλλωστε, δηλαδή υποστήριξη, ενίσχυση εισοδήματος με βάση τις ε, ανάγκες και την απόδοση. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει αυτή η, διά, διόρθωση του ΣΥΠΗΝ, δηλαδή η προσαρμογή του εισοδήματος ε, του γεωργού πάντα προσαρμόζεται, ε, ε, προσανατολίζεται σε αυτή την ενίσχυση, ενώ η γεωργική πολιτική θα πρέπει να επιδιώκει και την ανάπτυξη της υπαίθρου και όλα τα άλλα μέτρα, την οικολογικοποίηση, την προστασία της δημόσιας υγείας και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου λοιπόν εν ώψη και της μελλοντικής διαμόρφωσης μιας κοινή γεωργικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικό να πληρούνται και οι όροι του δεύτερου πυλώνα. Και πρέπει να κάνουμε τις αναλύσεις με βάση κάθε έκθεση που έρχεται ε, εάν έχουν υλοποιηθεί οι όροι και βεβαίως εάν υπάρχει περιθώριο για περικοπές στην περίπτωση των πρημοδοτήσεων αυτών και θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο, αν μπορεί να υπάρξει κάποιο ανώτατο όριο. Και με τον τρόπο αυτό να αποκλείσουμε για το μέλλον πιθανές εθνικές αξιολογήσεις για αυτές τις ε, ε, ε ενισχύσεις. Και ρωτώ ποιος ίσως να θεωρείται υπέτειος θα είναι η Περιτροπή, θα είναι τα κράτη-μέλη για, για τον κακό επιμερισμό των κονδυλίων, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Σε τελευταία ανάλυση έχουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία βεβαίω θα πρέπει να ε, διανέμονται στους δικαιούχους με βάση τα τα δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και τα κράτη-μέλη όπως και το ελεγκτικό συνεδρίο να μεριμνούν ώστε να γίνεται σωστή χρήση των κονδυλίων αυτών που προέρχονται από την τσέπη του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Άρα πρέπει να βρούμε ε, τη λεπτή αυτή ισορροπία και της ε, διάθεσης με το σωστό τρόπο του επιμερισμού, με σωστό τρόπο των κονδυλίων, αλλά και ταυτόχρονα της αποφυγής επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης κατά τον επιμερισμό αυτό. Μιλούμε βέβαια για απλοποίηση και την υποστηρίζουμε πάντα, αλλά αυτό δεν μπορεί να, σημαίνει, ότι δεν θα γίνεται σωστά η κατανομή, γιατί πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες. Και αυτή η ανάλυση των αναγκών για κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητη και πολύ σύντομα. Κλίντς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπαν και οι δύο προηγούμενες το θέμα είναι εδώ ε, ένα κεφάλαιο του προπολογισμού με τεράστια αντίκτυπο 18 δισεκατομμύρια το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι στόχοι που τύφονται και συνδέονται με το κονδύλιο αυτό να επιτυχάνονται. Για τους στόχους αυτούς ε, συμφωνούμε, νομίζω. Σωστή παραγωγή τροφίμων, σωστή, ε, σωστό εισόδημα για τους ε, Γιώργος. Όλα αυτά μας βρίσκουν σύμφωνους. Να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια και τον ε, υπεύθυνο του ελεκτικού συνεδρίου που μας παρουσίασε τα στοιχεία αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι πολλά τα ανοιχτά και τα εκκρεμή ακόμα ζητήματα. Το ελεκτικό συνέδριο γενικά ε, παρουσιάζει τα θέματα κριτικής με πολύ μεγάλη ευγένεια, αλλά έχει πολλά να θίξει στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε και η κυρία Κλάουντα Σμιτ και η κυρία Κάνιμπαχ. Εμείς ως ε, εισηγητές του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε κατά πόσον θεωρούμε ότι υπαρκούν οι εξηγήσει αυτέ του ελεκτικού συνεδρίου, όσο καλέ και να είναι ποιοτικά, ή μήπω χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι σε τέτοια μεγέθη θα πρέπει να εξετάσουμε μήπω θα πρέπει να κάνουμε και πιο πολλά από αυτά που κάνουμε στην παρούσα φάση γιατί είναι πολύ, και κρίσιμη, πολύ κρίσιμη και η χρονική συγκυρία. Σύντομα θα οριστεί το επόμενο στο πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η σωστή χρονική στιγμή να διορθώσουμε τα προβλήματα. Αν σωστά λοιπόν κατάλαβα η σύμπραξη μεταξύ ε, Ευρωπαϊκών ε, Κρατών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ε, απόλυτα όμαλη. Θέλουμε επικουρικότητα. Αλλά εδώ δεν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ του τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Ή το περιθώριο το οποίο έχει δοθεί στα κράτη-μέλη τελικά έχει οδηγήσει σε μια κατακαιρματισμένη κατάσταση. Και τελικά τι προκύπτει από τον ενεργό γεωργό και τον όρο αυτό. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των 18 αυτό δισεκατομμυρίων. Και όχι επειδή τα κράτη-μέλη εκμεταλλεύονται με διαφορετικό τρόπο το περιθώριο που τους δίνεται, τελικά να καταλήγουμε σε διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικά δικαιώματα. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Το ερώτημα για το κατά πόσον η έκταση των καλλιεργειών ε, θέλουμε να αποτελεί βασικό κριτήριο ή κατά πόσον υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θεωρούμε ότι είναι πιο κατάλληλα. Και αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε ως ερώτημα. Γιατί σε τελική ανάλυση θέλουμε να αλλάξουμε την ποιότητα της γεωργίας και το λέω αυτό όχι ως πράσινος, ως φιλελεύθερος το λέω αυτό. Θέλουμε να αλλάξουμε την εκτροφή θέλουμε να απομακρυνθούμε και να αφήσουμε πίσω μας ε, τη μαζική εκτροφή. Θέλουμε πιο βιολογικά και οικολογικά προϊόντα και παράλληλα θέλουμε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Το κατά πόσον αυτό συμβαίνει ήδη, πραγματικά θα το αμφισβητήσω. Το 2013 με τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, καταρτήσαμε έναν ε, αρνητικό κατάλογο, μια αρνητική λίστα για τις δραστηριότητε που δεν είναι κατ' ουσίαν γεωργικής ε, φύσεως. Από ό,τι κατανοώ, αυτή η αρνητική λίστα δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Μήπως να ελέγξουμε κατά πόσο θα επιμείνουμε ή μήπω να το καταργήσουμε πια αυτόν τον αρνητικό κατάλογο ή να αναπτύξουμε κριτήρια βάσει των οποίων οι ετούντε θα μπορέσουν να αποδεικνύουν καλύτερα το καθεστώ του ω ενεργοί γεωργοί. Τελευταίο σημείο. Το ερώτημα των τεσσάρων βασικών συστάσεων του Ρεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τη σωστή παροχή των επιφωτήσεων, τη διανομή πληροφοριών και το ρόλο των ε, οργανών πιστοποίησης. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια προσθήκη, μπορούμε να κάνουμε μια διόρθωση προκειμένου οι διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών αν δεν μπορούν να εξαλειφθούν τελείως, τουλάχιστον να μειωθούν. Σύντομα, λοιπόν, συντομία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σωστή η κατανομή των πόρων αυτών, προκειμένου αν υπάρχει τελικά αυτή η κοινή γερική πολιτική να έχει ως στόχο τη μείωση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έβαλα και τον εαυτό μου στην ημερήσια διάταξη, στην καταλάβη των ομιλητών, συγγνώμη. Πιστεύω, δεδομένου του περιεχομένου των, της έκθεσης, οι συστάσεις του κύριου Φιγκερέρα είναι εντελώς ανεπαρκείς. Είμαι πολύ απογοητευμένη, γιατί οι συστάσεις είναι πάρα πολύ αδύναμες σε σχέση με την έκθεση. Γιατί είναι τόσο αδύναμες λοιπόν και ανούσιες αυτές οι συστάσεις. Έχουμε διαβάσει την έκθεση και έχουμε κάτι κατά νου. Είμαστε κάπως ενήμεροι. Το θέμα είναι το εξή. Στην έκταση γίνονται πολύ βασικέ ε, διαπιστώσει και τα πορίσματα είναι σημαντικά. Σα ευχαριστώ. Αλλά τα συμπεράσματα, το τι θα κάνουμε με αυτά τα προβλήματα που έχουμε, πολύ απλά δεν αρκούν. Είχα φανταστεί κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει. Τα παραδείγματα τα οποία αναφέρεται μου άρεσαν πολύ. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό, όταν βλέπουμε ότι από 0,01 εκτάρια παίρνει κανείς ε, Ξέρουμε πόσο είναι το εκτάριο, 10.000 εκτάρια. 100 επί 100 λοιπόν τετραγωνικά μέτρα είναι το εκτάριο. Όταν έχω 0,01 εκτάριο έχω μια έκταση ενός το τετραγωνικό μέτρο. Σε αυτό το τετραγωνικό μέτρο δηλαδή 100 επί 100 παίρνω 9.000 ευρώ και παραπάνω. Μα ποιος θα μας... Ε, ποιος θα εγκρίνει αυτά. Αν το καταλάβει ο κόσμος και πει ότι «Α, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα φανταστεί έτσι την Ευρώπη σας», το καταλαβαίνω. Να ζητήσω λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμπεράσματα εξαγάγει. Μήπως κάποια πράγματα όχι μόνο που τα έχουμε σκεφτεί καλά, αλλά μήπως τα έχει περάσει και ελαφριά. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια τομή εδώ. Και θα ήθελα να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, τι συμπεράσματα βγάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από το συμπεράσμα ότι δεν θέλει να έχει να κάνει τίποτα με το θέμα αυτό. Γιατί τελικά με το μοντέλο αυτό ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και βγάζει όσο πιο πολλά γίνεται. Και το μοντέλο αυτό δεν μπορούμε να το πουλήσουμε ως πολιτική, γεωργική πολιτική. Και τελικά αυτή η ρήτρα ότι κρατήσετε τα χρήματα που δεν ξοδεύετε θα είναι πολύ αρνητική γιατί όλο και πιο λίγα θα είναι τα κρατημέλη τα οποία θα διαμορφώνουν ένα πραγματικά αποφατικό σύστημα. Άρα η έκθεση ήταν καλή. Οι συστάσεις ήταν πολύ αδυναμές. Και σκέφτηκα κι εγώ. Τι πρέπει να κάνουμε. Στα όρια της απόγνωσης είμαστε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τα σφάλματα αυτά. Πιο πολύ γραφειοκρατία, πιο πολλέ ρήτρε, πιο πολλοί κανόνε. Πολύ φοβάμαι ότι τελικά ούτε αυτό θα επιφέρει τα αποτελέσματα τα οποία χρειαζόμαστε. Να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά πάλι ο κ. Φιγκερέιδο. Ο κ. Πάσκου από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη έχει το λόγο. Και να μα πείτε ό,τι έχετε να μα πείτε. Μην διστάσετε. Έχετε χρόνο. Thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω διάφορα σχόλια για την έκθεση και μετά θα επανέλθω και στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσατε ε, μετά την εισαγωγή που έκανε και το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου όπως επίσης και από τον εισηγητή. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας, γιατί θέλω να εμβαθύνω στη συζήτηση αυτή, η οποία είναι η τρίτη, για τα ευρήματα αυτής της έκθεσης του Ελληνικτικού Συνεδρίου για το βασικό σύστημα ενίσχυσης και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας πως υπάρχουν θετικά στοιχεία για την έκθεση αυτή. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Συμπέρασμα της έκθεσης είναι πως η δράση και απόδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οικοδόμηση αυτού του συστήματος στήριξης εισοδήματος του ε, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαίου ε, Γεωργού, 4 εκατομμύρια γεωργοί. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, εμείς έχουμε επαρκώς στηρίξει την εισαγωγή αυτού του βασικού συστήματος ενισχύσεων και έχουμε παρακολουθήσει επαρκώς τη διαδικασία εφαρμογής. Έχουμε δώσει επαρκή κατεύθυνση και τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν θετικά. Όσοι διαβάσουν την έκθεση θα πρέπει να καταγράψουν πως η έκθεση γενικά είναι θετική για το βασικό σύστημα ενισχύσεων και για το ρόλο της Κομισιόν στο σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση αυτού του καθεστώτος. Το Ελληνικό Συνέδριο καταλήγει πως το σύστημα αυτό εισήχθη επιτυχώς από τα κράτη-μέλη και μιλάμε για ένα κλάδο ε, που έχει 8 εκατομμύρια ε, δικαιοχώς. Και αν δείτε ε, ε, τις άμεσες ενισχύσεις είναι πάνω από 7 εκατομμύρια δικαιούχοι, τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να πούμε πως χρειάστηκε να γίνει μεγάλη προσπάθεια και από τις εθνικές αρχές σε αυτά τα πλαίσια και η έκθεση καταλήγει πως τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό κατάφεραν να ελέξουν τον κίνδυνο αυτών των υπολογισμών και δεν επηρεάστηκαν από ουσιαστικό ε, ποσοστό σφάλματος ε, τα αποτελέσματα. Και θα πρέπει να πω πως οι συστάσεις, γιατί μιλήσαμε για τις συστάσεις, οι συστάσεις όταν όλες είναι σχετικές προ ε, προς την Κομισιόν ε, έχουν γίνει δεκτές. Και όπως είπαμε στο παρελθόν, δεν μπορούμε να προδικάσουμε αυτή τη στιγμή, θα το κάνουμε σε κάποιες επόμενε επόμενες εβδομάδες, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προδικάσουμε ποιοι θα είναι ε, αυτές οι συστάσεις, αλλά υπάρχει στόχευση, απλούστευση, σύγκληση όλα αυτά τα θέματα θα ε, βρεθούν ε, στην ε, νομοθετική πρόταση για τη μετά το 2020 περίοδο. Είναι λοιπόν σε καλή τροχιά το σύστημα και η επίπτωση στο, στη στόχευση, στην απλούστευση και στη σύγκληση αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένη. Και αυτά τα τρία στοιχεία είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση που δημοσίευσε για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας για την ΚΑΠ μετά το 2020. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω πως η πρόσφατη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον ε, του πολιετές πλαισίου δημοσιονομικών προοπτικών και για τις άμεσες ενισχύσεις, ε, πως θα αποτελέσουν αυτές ένα ε, συστατικό στοιχείο αυτών των προοπτικών, θα είναι πιο ευθυγραμμισμένες πιο ε, καλά στοχευμένες στο μέλλον και θα είναι πιο, ισορροπημένη η, πιο ισορροπημένος ο επιμερισμός αυτών των πληρωμών μεταξύ γεωργών, μεταξύ κρατών μελών και αυτό θα το πετύχουμε σε κάποιο μέτρο με την εισαγωγή ενός ε, ε, υποχρεωτικού, μιας υποχρεωτικής οροφής ε, στο σύνολο των ενισχύσεων που πληρώνονται είτε με μια ε, σταδιακή μείωση των πληρωμών, ένα degressivity δηλαδή, έτσι ώστε οι μικρές και οι ε, ε, μισές εκμεταλλεύσεις να λαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των ενισχύσεων. Και για την κατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε και εκεί να έχουμε μία ε, σύγκληση έτσι ώστε να έχουμε πληρωμές οι οποίες θα είναι γύρω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο ευρύτερα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων προτείνουν ένα νέο μοντέλο παραδοτέων έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα με τους επιχειρηματικούς ε, στόχους ε, και σκοπούς και ένα νέο μοντέλο παραδοτέων που θα γίνει η πολιτική μας πιο απλή, πιο αποδοτική και παράλληλα πιο στοχευμένη μέσω ε, της αγωγής δύο στοιχείων Πρώτον, μεγαλύτερη επικουρικότητα, έτσι ώστε να έχουμε τα πολιτικά εργαλεία τα οποία προσαρμόζονται περισσότερο στις ανάγκες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Και δεύτερον, με μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε αποτελέσματα και όχι σε επίπεδο συμμόρφωσης με κανόνες που έχουν τοποθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν επιστρέψουμε, θα ήθελα να μιλήσω και για κάποια από τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τις επικρίσεις που ακούσαμε και για τη στόχευση ε, και για την απλούστευση και για τη σύγκληση. Θα ήθελα να σας πω πως είναι ξεκάθαρο πως το διοικητικό βάρος έχει αυξηθεί αρκετά με την τρέχουσα ΚΑΠ σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά θα ήθελα να σας πω πως η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο αυτό συμπεριλάμβανε πολύ λιγότερες εναλλακτικέ λύσεις για διαχείριση του βασικού συστήματος ενισχύσεων και αυτή η πρόταση θα είχε οδηγήσει κατά τη γνώμη μας σε ένα πολύ πιο απλό σύστημα στήριξης εισοδήματος των ε, γεωργών αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνομοθεσίας προστέθηκαν πάρα πολλά στοιχεία που έδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει μία ε, πιο ε, καθετμημένη προσέγγιση η οποία οδήγησε σε περίπλοκους κανόνες σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό ε, για τη διαχείριση και τον έλεγχο. Μιλήσαμε για αρνητικό κατάλογο, μιλήσαμε για την ρήτρα ε, κενής εκμετάλλευσης Όλα αυτά οδήγησαν σε ένα κανόνα που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αποτελεσματικός, αλλά επίσης αύξησε και το διοικητικό βάρος σε πολλά κράτη-μέλη. Για τη στόχευση, πιστεύω πως η έλλειψη στόχευσης που έχουμε στην έκθεση θα πρέπει να στοχεύουν τη στήριξη στους ενεργούς γεωργούς στα κράτη-μέλη, δηλαδή σε γεωργούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτογενή παραγωγή. Επίσης, τα κράτη-μέλη μπορούν να πετύχουν την στόχευση με διαφορετική κατανομή των ε, ενισχύσεων, μπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο και με στόχευση μεγαλύτερη του συστήματος στήριξης εισοδήματος των γεωργών, όχι μέσω του καθεστώτος βασικών ενισχύσεων, αλλά μέσω των άλλων καθεστώτων γιατί το βασικό σύστημα είναι μόνο το 50 με 60% των συνολικών άμεσων ενισχύσεων που δίδονται στα κράτη-μέλη για να πληρωθούν στους γεωργούς. Έχουμε τους μικρούς γεωργούς, έχουμε την συνδεδεμένη στήριξη, έχουμε τους νέους γεωργούς, έχουμε πολλά καθεστώτα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να στοχεύσουν καλύτερα τη στήριξη εισοδήματος για τους γεωργούς οι οποίοι ε, εξαρτώνται από αυτήν. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα η στόχευση να βελτιωθεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατατόπου ανάγκες των γεωργών. Να προσθέσω δε ότι έχουμε με ένα συγκεκριμένο ε, ιδιάζον χαρακτηριστικό του κλάδου της γεωργίας είναι η μεγάλη κατάτμιση. Μίλησα για 4 εκατομμύρια δικαιούχους για το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, 7 εκατομμύρια για τι άμεσε ενισχύσεις, μεγάλη κατάτμιση και για να τους προσφέρουμε στήριξη εισοδήματο θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτού του, ε, αυτής βελτιωμένης στόχευσης και της ελαχιστοποίησης των, ε, του διοικητικού βάρους. Και είναι σαφές πως εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιτόπου συνθήκες και να δούμε πως τελικά αν τα κάνουμε όλα εμείς θα καταλήξουμε σε ένα ε, γραφειοκρατικό τέρας. Ξέρετε πως ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αλλά εδώ είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο πως θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ καλύτερης στόχευσης αφενός αλλά και της ανάγκης της μείωσης της ε, ε περιπλοκότητας και σε επίπεδο διοίκησης, αλλά και για τους γεωργούς, για τη σύγκληση. Να σας υπενθυμίσω πως η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ως στόχο να δώσει μια ενιαία ε, μοναδική αξία για το καθεστώς βασικών ενισχύσεων στα κράτη-μέλη μέχρι το 20 μέχρι το 2019 και είδαμε πως κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας συνομοθεσίας δόθηκαν κάποιες αναλλακτικές λύσεις. Οπότε τα κράτη-μέλη στιγμή έχουν τρεις αναλλακτικέ λύσεις για την εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλησης, δύο πλήρης ε, ε σύγκληση, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα και μια τρίτη εναλλακτική που είναι η μερική σύγκληση, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι το 2019 σε κάποια κράτη-μέλη θα υπάρχουν ακόμα διαφορές στις αξίες των δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω και για το λεκτικό μας έργο δύο λόγια, που αποτελεί ένα από τα βασικά του, της έκθεσης και θα ξεκινήσω με το ποσοστό στο οποίο κατέληξε το ελεγκτικό συνέδριο για την βασική αξία ενισχύσεων και νομίζω ότι και τα δικά μας στοιχεία είναι τα ίδια με αυτό το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, στις διαδικασίες εκαθάρισης και συμμόρφωσης ακολουθούμε αυτά τα ποσοστά και δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη, οπότε αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει το θέμα που ε, τίθεται στην έκθεση και θα το παρακολουθήσουμε στα πλαίσια της διαδικασίας εκαθάρισης και συμμόρφωσης. Το Ελληνικό Συνέδριο επίσης θεωρεί πως οι φορείς πιστοποίησης θα να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο τη στιγμή που ελέγχουν τη δημιουργία των δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει το ίδιο και πιστεύουμε πως οι φορείς πιστοποίησης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτούς τους ελέγχους και αυτό ήδη βρίσκεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε με το συμπέρασμα του ε, Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεχόμαστε και τη σύσταση της σχετική. Αυτά είναι η γενική απάντηση, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα συγκεκριμένα ερωτήματα, να σχολιάσω την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης του εισοδήματος των γεωργών και να σας πω πως αν υπάρχει ένας χώρος στο γεωργικό κλάδο που παρακολουθείται στενά, που αξιολογείται και αναλύεται, είναι η κατάσταση εισοδήματος. Το κάνουμε βασιζόμενοι σε μικροοικονομικές πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εξετάζουμε την εξέλιξη σε επίπεδο εισοδήματος ανά τύπο εκμετάλλευσης, ανά τύπο περιφέρειας κτλ. και σε επίπεδο κράτους μέλους. Και το κάνουμε ε, μέσω του δικτύου για τα λογιστικά στοιχεία εκμεταλλεύσεων και το κάνουμε και σε μικροεπίπεδο ε, χρησιμοποιώντας ε, τα στοιχεία που μας προσφέρει η Eurostat. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρίσκεται το εισόδημα το οποίο ε, γεννά η γεωργική δραστηριότητα στις εκμεταλλεύσεις αλλά και το εισόδημα που προκύπτουν από τη χρήση ε, των παραγωγικών μεσών ε, της εκμετάλλευσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, αγροτουρισμός ή πρώτη μεταποίηση επί της εκμετάλλευσης κάποιων προϊόντων. Οπότε ναι, αναλύουμε την κατάσταση εισοδήματο και αυτές τις πληροφορίες τις λαμβάνουμε υπόψη πρώτα απ' όλα για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη καθεστώτος στήριξης εισοδήματο. γιατί είναι μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού της ΚΑΠ και του ευρωπαϊκού προπολογισμού και νομίζω ότι εκεί έχουμε καλή τεκμηρίωση και επίσης χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές σε επίπεδο κρατών μελών για να γίνει και εκεί η καλύτερη ε, κατανομή και εξειδίκευση της κατανομής υπό την προϋπόθεση βέβαια πως δεν μπορεί να γίνει και εξατομίκευση αυτής της στήριξη. Είναι υπερβολικά ήδη και όχι στο γεωργικό κλάδο και δεν είναι παρόμοιος με άλλους οικονομικούς ε, κλάδους. Στήριξη εισοδήματο, χορήγηση αυτού. Το σύστημα για το βασικό καθεστώ ενίσχυση, που είναι ε, εκτατική ενίσχυση κυρίω. Και πρέπει να πω πως είναι σημαντικό για μας να διατηρήσουμε το εργαλείο αυτό ως εκτατικό εργαλείο. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ε, ένα από τα πιο αξιόπιστα, αξιόπιστες ε, πηγές πληροφόρησης και ο ΟΣΔΕ και ε, το σύστημα αναγνώρισης ε, αγροτεμαχίων. Έχουμε αναγνωρίσει εκατομμύρια ε, αγροτεμάχια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης είναι η πιο παραδοσιακή μορφή παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Είναι ο παράγοντας γεωργικής παραγωγής που απηχεί κατά τη γνώμη μας καλύτερα την, τον διοικό χαρακτήρα που είναι η παραγωγή τροφίμων αλλά και διαχείριση φυσικών πόρων και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Και με τον τρόπο αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε ένα σύστημα στήριξης εισοδήματος που θα βασίζεται στην έκταση. Και εδώ υπάρχει πολύ στενός συσχετισμός ε, με την κατανομή που γίνεται ε, με το βασικό καθεστώς ενίσχυσης, με τις πληρωμές εκμεταλλεύσεις και με το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Και γι' αυτό στην τρέχουσα περίοδο, και θα συνεχίσουμε κατά τη γνώμη μου, με την εισαγωγή μηχανισμών οι οποίοι προσπαθούν να απαλύνουν τις επιπτώσεις που έχει η μορφολογία του εδάφους και τα διαφορετικά μεγέθη των αγροτομαχίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον αρνητικό κατάλογο είναι ένα στοιχείο και αναφέρομαι εδώ στον ενεργό Γιώργο, για ένα στοιχείο που μπήκε στην νομοθεσία το 12 και το 13 με κάποιες τροποποιήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της χρήσης του αρνητικού καταλόγου για αδρανείς εκμεταλλεύσεις στην τρέχουσα ΚΑΠ και το ίμιση των κρατών μελών αποφάσισαν να αναστείλουν τη χρήση του αρνητικού καταλόγου και αντίστοιχα να χρησιμοποιήσουν από το 2018 τη ρήτρα ενεργής εκμετάλλευσης ενεργού γεωργού. Αυτό θα μειώσει και το διοικητικό βάρος και είναι προφανώς πως το παρελθόν τα πλειοψηφία των κρατών μελών έδειξε μία ε, επιθυμία να στοχεύσει την δημόσια ενίσχυση και κυρίως τη στήριξη εισοδήματο στους πραγματικού γεωργούς, δηλαδή οικονομικούς φορείς οι οποίοι παράγουν ε, εισόδημα μέσω γεωργικής δραστηριότητας. Για το παράδειγμα που δώσατε εσείς κυρία Πρόεδρε, για τη συγκέντρωση ε, της ε, ενίσχυσης μας σε πολύ μικρά αγροτεμάχια, να σας πω ότι υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει για το μέγεθος, για να μπορεί κανείς να λάβει αυτή την ενίσχυση και η σε θεμάχιο αναφοράς ε, είναι διαφορετικό από κράτος μέλος κράτος μέλος γιατί είναι διαφορετική διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων και του γεωργικού. 0,1 εκτάριο, δηλαδή ένα στρέμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο Και αυτό και για τις ε, μόνιμες καλλιέργειες και για την ανθοκομία ε, και για άλλες ε, πράσινες καλλιέργειες είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ελάχιστη απέτηση τεμαχίου το οποίο μπορεί να λάβει χρηματική ενίσχυση εισοδηματική. Και εδώ θα επιμένω υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές προϋποθέσεις όπου ο δικαιούχος θα προσπαθήσει να παρακάμψει τους κανόνες και να μεγιστοποιήσει τα εισοδήματα τα οποία, και τις ενισχύσεις οποίες λαμβάνει βάσει των δικαιωμάτων του και να σας πω πως οι δικαιούχοι αυτοί και πάλι υπόκεινται σε κυρώσεις από τα κράτη-μέλη, δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις υπερβολικής σώρευσης ε, ενισχύσεων, όπως επίσης και το θέμα της εσωτερικής ε, σύγκλησης μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα και ο Γιώργος αυτός θα αντιμετωπίσει αυτή την αποκλιμακούμενη ε, πληρωμή ενίσχυσης με τη σταδιακή κατάργηση που έχει φτάσει το 5% και σε νέα κράτη-μέλη έχουμε και οροφές στις ενισχύσεις που πληρώνονται στις γεωργούς. Οπότε έχουμε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν, πρέπει να το πω. Θα προσπαθήσουμε να τις αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον όπως κάνουμε σήμερα, αλλά θέλω να σας πω, προσέξτε. Είναι δύσκολο σε επίπεδο χάραξης πολιτικής να γενικεύει κανείς ότι πρέπει να γίνει ε, με βάση υποθέσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι πραγματικά κατεξαίρεση και που δεν υπάρχουν στη μεγάλη πλειοψηφία των γεωργών που λαμβάνουν αυτή την ισοδηματική στήριξη. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στόσο σε αυτό το θέμα. Οι εξαιρέσει. λέω ότι δεν εφαρμόζονται στο ίμιση τουλάχιστον το, οι εξαιρέσει με τι έκτακτες ρυθμίσει, αλλά αυτό σημαίνει ότι στι άλλε μισέ εφαρμόζεται. Και το βλέπουμε και από το έγγραφο και θέλω να ρωτήσω αν αυτή είναι η πρακτική, η πάγια πρακτική. Και δεύτερον, τι αλλάζει τώρα με τις ε, πρημοδοτήσεις με την έκθεση στην πράξη και για το προσεχές δημοσιονομικό έτος. Θα δούμε δηλαδή έκθεση για την οικολογικοποίηση και τους νέους γεωργούς μόνο χωρίς να αλλάξει τίποτε, δηλαδή ή θα αλλάξει κάτι. Τι αλλάζει στην πράξη, στην πραγματικότητα στην εκτέλεση της πρημοδότησης για νέους γεωργούς μέσα από την έκθεση. Και ευχαριστώ που μας δώσατε τόσο χρόνο. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε και εσείς ήταν δύσκολο να σας δώσω πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα είναι στη διαδικασία ε, προετοιμασίας και έγκριση συγκεκριμένη πρόταση για το μέλλον τη ΚΑΠ και είναι προφανέ πως η πρόταση αυτή θα περάσει και από τη διαδικασία συνομοθεσίας. Αυτό το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί στα πλαίσια τη ανακοίνωση για το μέλλον τη ΚΑΠ μετά το 2020 είναι η εισαγωγή ενός νέου μοντέλου παραδοτέων, που είναι πολύ σημαντικό για μας, όταν μιλάμε για απλούστευση, όταν μιλάμε για έλλειψη στόχευσης, όταν μιλάμε για έλλειψη αποτελεσματικότητας, δεν θα έλεγα αποδοτικότητας, γιατί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αποτελεσματικά αποδοτικό, και νομίζω ότι το ίμιση του εισοδήματο των γεωργών προέρχεται από την ενίσχυση και τη στήριξη εισοδήματο. Οπότε δεν νομίζω ότι εκεί έχουμε θέμα. Αλλά μπορούμε ε, σε κάποιο επίπεδο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί με ένα νέο σύστημα διακυβέρνηση, νέα παραδοτέα, έτσι ώστε να υπάρχει δημόσια ενίσχυση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους που θα θέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά οι οποίοι θα μεταφέρονται και θα ερμηνεύονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο βάσει των αναγκών που έχει εντοπίσει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο το κράτος μέλους και βάσει μια σειρά κανόνων που θα είναι απόλυτα σχεδιασμένοι από τα κράτη-μέλη βάσει ενός ευρωπαϊκού πλαισίου και που θα έχουν εξειδικευτεί πάνω στις ανάγκες των κρατών μελών έτσι ώστε η μελλοντική στήριξη εισοδήματο να είναι πολύ πιο προσαρμοσμένη, πολύ πιο εξειδικευμένη στις ανάγκες έτσι ώστε οι μικρές και μεσές εκμεταλλεύσεις να στηριχθούν περισσότερο και να μειωθεί η παροχή ενίσχυσης στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες, όχι αυτομάτως βέβαια, αλλά πολύ πιθανό, χρειάζονται λιγότερη δημόσια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι, κατά τη γνώμη μας, η βασική αλλαγή για το μέλλον. Μία αλλαγή ε, της, ε, του σκεπτικού που ακολουθούμε και για τη στόχευση να σας πω πως η στόχευση θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε το βαθμό απλούστευσης, θα μειώσει το πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα και όταν μιλάμε για τον αρνητικό κατάλογο, οι αρνητικοί κατάλογοι συντάχθηκαν στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως για πολλά κρατημέλη δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Οπότε στόχος μας θα είναι να στοχεύσουμε στους ενεργούς γεωργούς, πραγματικούς γεωργούς και ας ορίσουν τα κράτη-μέλη τι κατά τη γνώμη τους και σύμφωνα με τους δικούς τους κλάδους ποιος είναι ενεργός γεωργός. To the current situation, so we have a system which is Κάτι πιο απλό λοιπόν και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε είναι η εισαγωγή ενό πιο δικαίου συστήματος κατανομής στήριξη εισοδήματο για όλους τους γεωργού κάποιας χώρας και βέβαια σε επίπεδο κρατών μελών. Και αυτά στα πλαίσια του πολιετούς προγρα... πλαισίου. Μια και σας είπα πως για το μέλλον θα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα, αλλά η εφαρμογή αυτής της στήριξης θα γίνει με ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα έτσι ώστε να έχουμε πιο δίκαιη κατανομή. Και θα εφαρμόσουμε είτε σύστημα με οροφές, σε χαμηλά σχετικά ύψους. Νομίζω αυτή τη στιγμή ε, ε, σχεδιάζουμε, είτε ε, κλιμακωτή μείωση των πληρωμών που γίνονται σε εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να πληρώνονται περισσότερο οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ε, ε, περισσότερες ανάγκες μικρές μεσαίες εκμεταλλεύσεις και όχι πολύ μεγάλες. Που δεν χρειάζονται τόσο πολύ στήριξη. Αυτά. Νομίζω θα εγκριθεί σε επόμενες εβδομάδες αυτή η πρόταση και θα έχετε και πολλές λεπτομέρειες για το μέλλον της στήριξης Δήματος και του βασικού συστήματος ενισχύσεων ε, για την ΚΑΠ μετά το 2020 και αυτά θα τα έχετε σε μερικές εβδομάδες. Yeah, ναι, ευχαριστώ πολύ. Τα περιμένουμε με αδημονία. Και σημειώνω ότι δεν αλλάζει τίποτα προς την ε, νομική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Παραμένουν τα πράγματα όπως είναι, απλώς μπορεί μετά να βελτιωθούν. Η κυρία Κάντενμπαχ πρώτα, πρώτα ο κύριος του. Παρακαλώ. Ναι, στην παρουσίαση της ανακοίνωσης. Αυτό το νέο μοντέλο, το New Delivery Model, καλύπτει υποτίθεται το πρόβλημα πάνω στο οποίο συζητήσαμε, αλλά δική μου εκτίμηση τώρα αυτό προσωπική. Θεωρώ ότι όταν έχουμε μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν καταστάσεις, θα έπρεπε και να αναπτύσσει περισσότερες ε, δυνατότητες για αντικειμενικό και αξιολόγηση αυτή τη νέα κατάσταση που θα διαμορφώνεται με τη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε δηλαδή τι γίνεται. Και άρα χρειαζόμαστε δείκτε, παραμέτρου που θα εξασφαλίζουν συγκρίσιμη κατάσταση για τα διαφορετικά μοντέλα, σύγκριση μεταξύ των διαφόρων μοντέλων, αλλά και ταυτόχρονα μια δυνατότητα παρακολούθηση των εξελίξεων. νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση με διαφορετικά μοντέλα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα για την ε, αξιολόγηση με παραμέτρους. Και επίσης το ελεγκτικό συνέδριο. Σε ποιο βαθμό μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα κριτήρια για την ε, έκθεσή του, για τις εκτιμήσεις του. Άλλα σχόλια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ένα ζήτημα που έθεσε η κυρία Κάντενμπαχ. Στο μέλλον, εάν και νομίζω ότι είναι πολύ συμφωνές και προτάσεις Επιτροπής σε σχέση με τον σωλείο κανονισμός, θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο σχεδιασμού και εφαρμογής των κρατών μελών, από πλευρά των κρατών μελών, των ε, σχεδίων στήριξης, αλλά υπογραμμίζω αυτό θα γίνεται μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συγκεκριμένο. Δεν θα είναι ε, λευκό επιταγή. Θα υπάρχουν όροι, θα υπάρχουν προϋποθέσεις βεβαίως. Αυτό επεξεργαζόμαστε τώρα, το επίπεδο της λεπτομέρειας αυτών των μέσων, ακόμα δεν ε, έχει προσδιοριστεί το γενικότερο πλαίσιο. Τα κράτη από εκεί και πέρα θα μπορούν να βρουν τις ε, συγκεκριμένες λύσεις για να διαμορφώσουν τα έργα, τα προγράμματα που θέλουν, ε, τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να στηρίξουν ένα συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή κτλ. Αλλά δεν θα περιοριστεί ο γενικός στόχος. Αυτό γιατί, γιατί με το πρασίνισμα Φερρυπίνη, αν πούμε ε, για όλους ισχύουν τα ίδια ποσοστά, ε, δεν, ε, δεν μπορεί να ισχύουν και όλους τα ίδια ποσοστά γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες. Και έτσι εδώ θα μπορεί το να, το κράτος μέλος να προσδιορίσει τι θέλει. Μπορεί να μου πείτε θα είναι 27 διαφορετικά μοντέλα. Μα ούτως ή άλλως έχουμε διαφορετικά μοντέλα. Κοιτάξτε τώρα ποια είναι η κατάσταση αν που όπως έχει δημοφωθεί. Θα έχουν όμως μια πλαισίωση, ακόμα και 27 άρα τα νέα κράτη, θα έχουν μια πλαισίωση με επαρκή ευελιξία ώστε να ε, εξασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος της ενίσχυσης εισοδήματος και ο σχεδιασμός με βάση και τα όσα ζητεί το ελεκτικό συνέδριο, θα είναι ε, ένα σχεδιασμός με βάση καλύτερους στόχους, πιο συγκεκριμένους στόχους, αλλά και όχι μόνο στην υποστήριξη, στην ενίσχυση και στην ε, εξυπηρέτηση των κλιματικών προϋποθέσεων και όλα αυτά που προβλέπονται και για να επιτρέψει μια καλύτερη αξιολόγηση με ένα σύστημα αξιολογήσεων του αντικτύπου που θα έχουν τα διάφορα, μέλη, ε, τα διάφορα προγράμματα ε, ή τα μέτρα καλύτερα των ε, κρατών. Μετά το 2021 θα έχουμε δηλαδή μετρήσιμους δείκτες για να μπορούμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την κατάσταση. Με λίγα λόγια έχετε απόλυτο δίκαιο αγαπητοί συναδελφοί. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριος Φιγκερίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας αγαπητά μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις που κάνατε. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας για την έκθεση ελέγχου. Είπατε κάποιες γενικές, κάποια γενικά λόγια. Να πω καταρχάς λοιπόν κάποια γενικά λόγια. Φυσικά το ολεκτικό συνέδριο θα πρέπει να δίνει μια ομοιόμορφη άποψη όταν παίρνει το λόγο, αλλά θα πρέπει να είναι και σαφέ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι ξεκάθαρο. Πιστεύω λοιπόν στην έκθεσή μα. Ήμασταν ξεκάθαροι στο βασικό μήνυμα το οποίο μεταβιβάσαμε. Αλλά το να υπάρχει σαφήνεια σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρονική συγκυρία. Την εκάστοτε. Στην παρούσα λοιπόν φάση γίνονται μεγάλες συζητήσεις ε, για τη νέα οικονομική περίοδο, για τη νέα πολιτές πλαίσιο. Και θα πρέπει να είμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται δεδομένη της, της χρονικής συγκυρίας. Σε όλα τα ερωτήματα λοιπόν που έθεσες, που θέσατε, θα έλεγα ότι στην έκθεσή μας λέμε δύο πράγματα βασικά. Καταρχάς, ότι τυπικά το σύστημα είναι δρομολογημένο. Από τυπική άποψη είναι στο δρόμο. Αλλά επί της ουσίας ο βασικός στόχος, τα βασικά αποτελέσματα της ε, μεταρρύθμισης του 2013, αυτά που θέλαμε να πετύχουμε δηλαδή, επί της ουσίας δεν τα έχουμε πετύχει. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, τη στόχευση και τη σύγκληση. επί της ουσίας. Δεν τα έχουμε πετύχει. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να μεταβιβάσουμε προς τον νομοθέτη. Να προσέξετε λοιπόν εδώ. Να δείξουμε λοιπόν και κάποια άλλα ζητήματα. Καταρχάς, το θέμα του διοικητικού άχθους. Ναι, είναι σαφές για όλους ότι η απλούστευση ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης του 2013. Πιστεύουμε και θεωρούσαμε ότι συμφωνούσε μαζί μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η περιπλοκή της μεταρρύθμισης επί της ουσίας της. Οι πολλαπλές δυνατότητες που δόθηκαν στα κράτη-μέλη και όλες οι λύσεις τελικά που επιλέξαν τα κρατημέλα τα κρατημέλη ήταν πιο περιπλοκή τελικά από ότι οι κανόνες που είχαν οριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Να θέσω λοιπόν μια ερώτηση, μια βασική ερώτηση. Είναι κακό να δίνουμε εξουσία στα κρατη να εφαρμόζουν συγκεκριμένες λύσεις. Πιστεύω πως όχι. Υπό έναν όρο όμως. Αν υπάρχει ένα γενικό κανόνας αν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη, το οποίο θα πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Αν δεν υπάρχει γενικό πλαίσιο, αν δεν υπάρχει γενικός κανόνας και δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι επιθυμούν, τι διαπιστώνουμε τελικά. Ότι οι τελικές λύσεις είναι πιο πολύ σύνθετες. Δεν υπάρχει απλούστευση. Και όπως είπε ο κύριος Βάσκου, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί μαζί μας από αυτού. Δεύτερη ερώτηση, την οποία θα ήθελα να κάνω. Διαφορές μεταξύ χωρών. Είναι τεράστιες ποσοτικά, σε ό,τι αφορά τα ποσά δηλαδή, που χορηγούνται. Συμφωνούμε και όπως ε, το βλέπετε και από την έκθεσή μας. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι γιατί. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στα ποσά Και εδώ θεωρώ ότι οι είναι... Η απάντηση είναι τριπλή. Καταρχάς, ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει ο νομοθετής. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των γεωργικών καταστάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι γεγονός και δεν αλλάζει εύκολα. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Έχουμε όμως δύο άλλους τομείς όπου ενδεχομένως ο νομοθέτης μπορεί να ε, παρέμβει. Καταρχάς, ε, το στοιχείο των ιστορικών ε, παραγόντων. Πιστεύω. Έχουμε ακόμα ένα ιστορικό βάρος πάνω μας. Έχουμε στοιχεία από την αρχή του αιώνα που προκαλούν διαφορές στα ποσά που καταβάλλονται στους αγρότες. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία θα πρέπει να κάτσει να τα εξετάσει ο νομοθέτης. Δεύτερο στοιχείο, οι δυνατότητες που έχουν δοθεί στα κρατημέλη για να χρησιμοποιήσουν όποια λύση επιθυμούν. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι καλό το ότι δίδεται διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Αν υπάρχει όμως ένας γενικός κανόνας, ένα γενικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Αυτά για τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Η τρίτη πτυχή στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ και την οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω, πολύ σημαντική για μας, η έλλειψη μιας ε, κοινή βάσης. Δεν υπάρχουν ε, επαρκείς κοινές βάσεις ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το εισόδημα των γεωργών. για να υποστηριχθεί επαρκώς και με ασφάλεια ο εκάστοτε στόχος της πολιτικής σε ό,τι αφορά την ε, προστασία, για παράδειγμα, του εισοδήματο των γεωργών. Δεν έχουμε κοινέ ε, τέτοιε βάσει. Μια κοινή γραμμή βάσεις. Και επίσης πιστεύουμε ότι η ελλείψη τέτοιων κοινών βάσεων στην τρέχουσα ΚΑΠ δεν υπάρχει και σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής, των πολιτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων αυτών και των ποσοτικών μέτρων. Καμία σύνδεση. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι ένα συγκεκριμένο πολιτικό εργαλείο ε, έχει αποτελεσματικότητα ή όχι. Γιατί δεν έχουμε γραμμές βάσης, δεν έχουμε προσωπικούς στόχους και δεν υπάρχει και σύνδεση μεταξύ των πολιτικών και των εργαλείων. Τέλος, το θέμα ε, των στόχων και της αρνητικής λίστας. Όπως το είπε ξεκάθαρα και ο κύριος Πάσκο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η ιδέα της αρνητικής ε, λίστας ε, την έθεσε το Κοινοβούλιο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν καλή ιδέα. Ήταν καλή ιδέα. Γιατί αυτός ο αρνητικός κατάλογος ουσιαστικά ήθελε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε. Μεγάλο μέρος της οικονομικής βοήθειας τελικά χορηγούταν σε ανθρώπους που δεν ήταν γεωργοί στην τελική ανάλυση, δεν ήταν αγρότες. Αυτό λοιπόν στην ήταν καλό. Αλλά τι διαπιστώσαμε τον των υστέρων, ότι αυτή η συγκεκριμένη λύση ευνόησε την περαιτέρω περιπλοκή του συστήματος και την περαιτέρω γραφειοκρατικό άχθος στα κράτη-μέλη. Και εδώ θα είμαι ξεκάθαρος. Θα σας πω το εξής. Τι λύση βρήκε το Κοινοβούλιο για τα προβλήματα αυτά. Η λύση, πολύ λυπάμαι που σας ενημερώνω και το λέω, αλλά το λέω με κάθε ε, πίστη προς το Κοινοβούλιο, ότι η λύση την οποία πήρε το Κοινοβούλιο ήταν η πιο εύκολη. Να πει ουσιαστικά στα κράτη-μέλη, κάντε ό,τι θέλετε. Το Κοινοβούλιο δεν ρώτησε γιατί έχει περιπλακεί τόσο πολύ γραφειοκρατικά η κατάσταση και τι λύσεις μπορούμε να βρούμε σε ό,τι αφορά τη στόχευση. Όχι. Το κοινοβούλιο πήρε την εύκολη λύση. Κάντε ό,τι νομίζετε. Χωρίς ένα γενικό κανόνα. Χωρίς ένα γενικό πλαίσιο. Γι' αυτό χαίρομαι που ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εισακούσουμε και μελλοντικέ προτάσει. Λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα δούμε τι λύσεις θα μας προτείνουν. Τέλος. Να πω το εξής. Συμφωνώ και να μην ξεχνάμε ότι στην γεωργική πολιτική Έχουμε τα καθεστώτα βασικών ενισχύσεων, έχουμε και όλες αυτές τις ανησυχίες για το εισόδημα των γεωργών, αλλά έχουμε και άλλες ανησυχίες. Περιβαλλοντική προστασία, δημόσια υγεία, ευημερία των ζώων. Έχουμε τόσους πολλούς παράγοντες να συνυπολογίσουμε. Και είναι πολλαπλές οι εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει το ελεκτικό συνέδριο για όλους αυτούς τους τομείς και είμαι βέβαια ότι είστε για να υπάρχει επισκόπηση των προβλημάτων που εμπεριέχονται εδώ στον τομέα της ε, γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τις συστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τα κρατικά σχόλια που έχετε να κάνετε για τις συστάσεις μας. Κατανοώ πώς αισθάνεστε. Αν πιστεύετε και ακούσετε όμως με προσοχή τι λέμε, οι συστάσεις στις οποίες προβήκαμε, λαμβάνουν υπόψη και την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ξεκινάμε μια νέα πολιτική και προβαίνουμε σε συστάσεις τους τρεις βασικούς τομείς που θεωρούμε τους πλέον σημαντικούς. Γιατί στο μέλλον θα βρούμε πολλές λύσεις ε, για το θέμα της ε, απλούστευσης, για το θέμα της στόχευσης, αλλά ποια είναι τα βασικά ζητήματα, τα πραγματικά ζητήματα. Καταρχάς, να προσέξουμε τις υπολογισμούς, γιατί αν θέλουμε να δώσουμε ενισχύσει στους γεωργούς για να κάνουν άμεσες υπολογισμού για μας, ο εξωτερικός έλεγχος είναι πολύ βασικό στοιχείο. Αυτό λέει ουσιαστικά από τη σύσταση. Δεύτερη σύσταση. Για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν καλές πληροφορίες σωστές πληροφορίες και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει επαρκείς πληροφορίε, όχι εγκαίρω, εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και γι' αυτό λοιπόν στη σύσταση υπαριθμών 2 ακριβώ αυτό τονίζουμε, το θέμα τη πληροφόρηση τη ενημέρωση. και πιστεύουμε και ζητάμε στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ακόμα πιο πολλέ αρμοδιότητε και ακόμα πιο πολλέ εξουσίε να ζητάει στοιχεία από τα κράτη-μέλη προκειμένου και Επιτροπή και Κοινοβούλιο να έχουν επαρκεί πληροφορίε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των πολιτικών. Τρίτη σύσταση τώρα. Το βασικό ζήτημα. Το κεντρικό ζήτημα που θεωρούμε ότι συνδέει πάντα. Έλλειψη κοινών γραμμών βάσεων, βάσης σε ό,τι αφορά το εισόδημα των γεωργών. Γιατί αν έχει ένα βασικό στόχο η γεωργική πολιτική που είναι η ενίσχυση του εισοδήματο των γεωργών, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχουν γραμμές βάσει για τους στόχου αυτούς, προκειμένου να υπάρχει σωστή στόχευση, προκειμένου να υπάρχει πραγματική και σωστή σύγκληση. Ελπίζω, Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής, να απάντησα στα πιο βασικά ζητήματα στα οποία και αναφερθήκατε, αλλά φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω και σε περαιτέρω ερωτήσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Also. Κυρία Πάντα μπορεί να πει κανεί πολλά, αλλά το να μιλάει, το να μονολογεί για πολλή ώρα δεν σημαίνει ότι δίνει και απαντήσεις ε, στα ζητήματα ή ότι εξυπηρετεί το στόχο. Είπα και εγώ ότι υποστηρίζω κάποιε από τις προτάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία, φορά, από τη μία πλευρά να καλείται το κοινοβούλιο και εμείς να προσπαθούμε μέσα από την Επιτροπή μας να υλοποιήσουμε ό,τι το καλύτερο και να ζητούμε με τι ε, ειδικέ εκθέσεις ακόμη περισσότερη διαφάνεια, σαφήνεια, πληροφορίε και μετά να μας κατηγορούν ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη αρκετά από τα στοιχεία αυτά. Δεν το δέχομαι αυτό. Είναι ακραίο και θεωρώ ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει περισσότερες εξουσίες. Άλλωστε είναι και βασική αρχή της ε, επικουρικότητας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι ε, ισχύει και πώς είναι δυνατόν μέσα από τις διαδικασίες να διευκολύνουμε και, να γίνεται, και, και τα κρατημέλη αλλά και να γίνεται η δουλειά καλύτερα στο επίπεδο που είναι καλύτερα γενομένη. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν. Όλα τα άλλα νομίζω ότι περιτεύουν. Ευχαριστώ, η Ούτω ή άλλω αυτό είναι ένα θέμα και το επισημένο που δεν θα το λύσουμε εμεί, αλλά η Επιτροπή Γεωργία, η οποία ορίζει και του κανόνε εν όλο που επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς. Η Επιτροπή μέσα από τους τριμερείς βιολόγους έχει βεβαίως πολλές δυνατότητες. Εάν δεν τις αξιοποιεί, ε, τι να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή να μας λέτε «Α, στην προσοχή μεταρρύθμιση, όπως έχουμε έχει ήδη συμβεί, θα τα καταφέρουμε καλύτερα» και πάλι να είναι η κατάσταση μη ικανοποιητική. Ε, εντάξει, δεν, ε, έχω περάσει τόσα χρόνια που περιμένω να γίνει καλύτερη κατάσταση, δεν θα παραιτηθώ τώρα. Καταλαβαίνω ότι επιδιώκει περισσότερες εξουσίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και το αντίστροφο, δηλαδή σπρώχνουν τα πάντα προς τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση και την αρχή της επικουρικότητας έχει ρόλο να εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως να φτάσω και σε αυτό, το ζήτημα των 20 μεγαλύτερων ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είπαμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά, μα εσείς από τις πληροφορίες που έχετε στη θέσή σα. είναι δυνατόν να μου λέτε ότι δεν έχετε στοιχεία. Δεν, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία και περίμενα μια πολύ συγκεκριμένη ανάλυση. Εάν δεν το κάνει η Επιτροπή, ποιος θα το κάνει. Εδώ έχουμε να κάνουμε τεράστια ποσά. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν σαμάνα εξ ουρανού σε όλη την Ευρώπη χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμούμε, να αξιολογούμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Και κύριε Φιγκέιρέντο, ελπίζω ότι θα, μπορέ, ότι θα έχετε ήδη, ότι θα μπορέσετε σύντομα, ναι, Ωραία, να παρουσιάσετε αυτή την ειδική έκθεση στην Επιτροπή Γεωργίας. Μάλιστα, έχετε και ορίσει και, για κουνήστε το κεφάλι να καταλάβω, ε, έχετε κανονίσει και ημερομηνία παρουσίασης. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Ολοκληρώσαμε εδώ αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συζήτηση. Ολοκληρώθηκε εδώ η, ε, το δημόσιο κομμάτι της συνεδρίασής μας. Όσοι δεν έχουν συνεργασία να αποχωρήσουν ησύχω και ταχαίως. Αλλιώς συνεχίζουμε το απόγευμα στις